Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν τελειώσει το πρώτο πάνελ. Να περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην πρώτη ακρόαση με τίτλο Οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τομεί δραστηριότητες ε, και μέσα πρόληψη, έρευνα και καταστολή. Καταρχήν ε, θα ακούσουμε τη UNDC και την Interpol που θα μας δώσουν μια γενική αξιολόγηση του οργανωμένου κλίματος σε παγκόσμιο Θα ξεκινήσουμε αμέσω ακούγοντας την κυρία Με, η οποία εκπροσωπεί το, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών ε, κατά του οργανωμένου εγκλήματος ε, και των ναρκωτικών και θα μας μιλήσει για την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διακίνηση των ναρκωτικών με μια συνθετική παρουσίαση της έκθεσης, της Παγκόσμιας Έκθεσης για τα Ναρκωτικά και θα μας κάνει και μια λεπτομερή ανάλυση σε παγκόσμιο επίπεδο για την ε, προσφορά την κατανάλωση και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Και κατόπιν θα έχουμε τον εκπρόσωπο της Ιντερπόλ, τον κύριο Ρόσμπαχ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια καθολική αξιολόγηση, παγκόσμια αξιολόγηση της οργάνωσής του σε σχέση με τις απειλές για το οργανωμένο έγκλημα. Σε σχέση τώρα με τον χρόνο, θα πρότεινα να οργανώσουμε ως εξή τη συζήτηση, να δώσουμε απευθεία στην κυρία Με, η οποία θα κάνει μια παρουσίαση 15 λεπτών και έκανα μια εισαγωγή. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το κάνω και καθώς την τελευταία φορά ε, είχαμε ε, ουσιαστικά κάπως υπερβεί τους χρόνους και τελικά κάποια στιγμή εγώ αναγκάζομαι να σταματήσω δορμηλητή Έτσι λοιπόν θα σας παρακαλώ να 15 λεπτά και ο κύριος Ζώσπαχ να μιλήσει για 15 λεπτά και τώρα και κατόπιν μάλλον θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θα το ζητήσουν. Και φυσικά ο εισηγητής και οι συντονιστές των ομάδων έχουν προτεραιότητα. Όταν υποβάλλετε τις ερωτήσεις θα ήθελα να σας πω, να μας λέτε με συγχωρείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας και να σας πω ότι έχουμε μόνο δύο λεπτά για τις ερωτήσεις κατόπιν θα απαντήσουν οι εισηγητές και αν υπάρχει ακόμη χρόνος στη διάθεσή μας θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων και έτσι θα μπορέσουν εκ νέου να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Τώρα, για να μην ε, χάσουμε άλλο χρόνο, κυρία με παρακαλώ. Eh, Καλημέρα σας, ε, κύριε Πρόεδρε αν ε, έχω φτάσει στα δύο τρία λεπτά πριν να τελειώσει η ομιλία, να μου, δώσετε, να μου κάνετε ένα σήμα. Λέγομαι Έτζελα Μέη, είμαι από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ορισμένα από τα κύρια απορίσματα της Παγκόσμιας Έκθεσης για τα Ναρκωτικά που δημοσιεύουμε κάθε έτος όπως μπορεί να γνωρίζετε και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει παγκόσμια στις αγορές ναρκωτικών. Θα προσπαθήσω να σας ε, παρουσιάσω ορισμένα από τα στοιχεία που αφορούν κυρίως την Ευρώπη και ορισμένες από τις αναδυόμενες τάσεις ε, που βλέπουμε ε, στην Ευρώπη αλλά και τις διαδρομές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, να σας πω τι βλέπουμε. Δεν βλέπουμε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τη χρήση των ναρκωτικών, αν δείτε εδώ τις μπάρες ε, και με το καφέ και με το μπλε, έχουμε εδώ τον καθολικό αριθμό ε, των χρηστών ναρκωτικών παγκοσμίω ε, και βλέπετε ότι δεν βλέπουμε ιδιαίτερε αλλαγές να σημειώνονται με την αλλαγή των ετών. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή δεν βλέπουμε μεγάλες παραγωγές στην παγκοσμία παραγωγή κοκαίνης, σε ό,τι αφορά την παραγωγή οποίου είδαμε ότι η παγκόσμια παραγωγή επέστρεψε για το οποίο περίπου στις 7.000 κυβικούς τόνους ε, που παράχθηκαν το 2011 μετά από μία πτώση που είδαμε το 2010 ε, λόγω μιας νόσου που έπληξε τα φυτά του οποίου στο Αφγανιστάν ε, και μειώθηκαν οι εισοδιές στο Αφγανιστάν κατά περίπου 50%. Και βλέπουμε κάποιες αλλαγές ε, και να σας ε, να σας πω να δούμε την ε, διακίνηση της ηρωίνης. Η ηρωίνη προέρχεται από το Αφγανιστάν, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, αριστερά. Φεύγει από το Αφγανιστάν, περνά από το Ιράν, την Τουρκία και τα Βαλκάνια και φτάνει στη Δυτική Ευρώπη και υπάρχει και η Βόρεια Οδός μέσω της Κεντρικής Ασίας ε, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτές είναι οι δύο κυρίες αγορές καταναλωτών που βλέπουμε. Υπάρχουν ε, και άλλες οδοί, γιατί βλέπουμε τώρα το αφγανικό όπιο να πηγαίνει και προς τα νοτιοανατολικά, αλλά αν θέλουμε να επικεντρωθούμε ιδίω στη Δυτική Ευρώπη, βλέπουμε αυτή την παραδοσιακή οδό. Τι βλέπουμε λοιπόν δείτε εδώ. Αν δείτε εδώ ένα χάρτη, Βλέπουμε αποστολές ηρωίνη από το Αφγανιστάν που να φτάνει στο Πακιστάν και μέσω τη ε, θάλασσα για τη ε, πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Κατάρ. Και κατόπιν ε, διασύζει τον κόλπο για να κατευθυνθεί στην Ανατολική Αφρική. Τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες κατασχέσεις ε, στην Ανατολική Αφρική που αυξήθηκαν κατά 200%. Και πάλι εξακολουθεί να παραμένει μικρό το ποσοστό, αλλά βλέπουμε μία οδό που επεκτείνεται. Και τι βλέπουμε, ιδίως ότι η ηρωίνη που συνήθως ερχόταν οδικά στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες αγορές, ε, τώρα έρχεται μέσω ε, κάποιων ε, κόμβων και εμπορικών οδών, όπως είναι το λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα. Γίνεται πραγματικά κόμβος για τα για την εμπορία των αγαθών. Και φυσικά ε, η αγορά τη ηρωίνη εκμεταλλεύεται αυτό το μεγάλο αριθμό κοντέινερ και ε, επιβατικών αεροπλάνων που περνούν ε, από το Κατάρ και από τα Ηνωμένα Ναυικά Εμμυράτα και βλέπετε σε αυτό το τμήμα του κόλπου να αναδύεται ένας κόμβος και για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Βλέπουμε την ηρωίνη από το Πακιστάν να περνά στα Ηνωμένα Βελικά και να επιστρέφει στην Κίνα, αλλά και απευθεία στην Ευρώπη. Και με το αεροπλάνο, αλλά και τη θαλάσσια οδού. Η Ισπανία το 2011, πριν το ανέφερε μια αύξηση περίπου 15% των κατασχέσεων στα λιμάνια, ενώ πριν μάλλον το, ε, σχεδόν το 50% των κατασχέσεων που είχαν ε, για την ηρωίνη ήταν στα λιμάνια, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν αμελητές αυτές οι κατασχέσεις. Έτσι λοιπόν η ηρωίνη φτάνει στην Ευρώπη και για τις θαλάσσιες οδού. Αν ε, δούμε τώρα τι συνέβη το 2010, υπήρξε αυτή η ασθένεια των φυτών, όπως σας είπα, στο Αφγανιστάν, και μειώθηκε δραστικά η παραγωγή της ηρωίνης. Και τι είδαμε. Πώς μεταφράστηκε αυτό στην αγορά της Ευρώπης. Σε αυτό το χάρτη βλέπετε με μπλε τις κατασχέσεις. Εδώ βλέπετε τις κατασχέσεις και με το μπλε βλέπετε ότι υπάρχει μείωση των κατασχέσεων. Ενώ με το καφέ βλέπετε που υπάρχει αύξηση. Ενώ η κίτρινη φυσαλίδα σημαίνει ότι υπάρχει σταθερότητα στην Κίνα, παραδείγματο χάρη. Και όταν ε, είχαμε αυτή την νόηση των φυτών στον Αφγανιστάν, μέσω όλες αυτές τις οδού που σα έδειξα πριν από το Αφγανιστάν προ τη Δυτική Ευρώπη, είδαμε μία μείωση στι κατασχέσει. Και καθώ ε, αυτό συνέβη, καθ' όλο το μήκο τη οδού, αυτό μα δείχνει ότι υπήρξε μείωση της ε, προσφοράς ηρωίνης. Επίσης, ε, έχουμε κάποιες ενδείξεις ε, για έλλειψη ηρωίνης σε κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εκεί μπορεί να υπάρχει ένα συνδυασμό καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο, η ηρωίνη μάλλον που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποστέλλεται απευθεία από το Πακιστάν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότεροι ηρωίνοι δηλαδή δεν ακολουθούν την οδό που σας έδειξα πριν, και υπάρχει άμεση επίπτωση από την έλλειψη οποίου στο Αφγανιστάν. Και υπήρξε λοιπόν έλλειψη ηρωίνης ε, στην αγορά ηρωίνης και μπορεί να οφείλεται όχι μόνο στην ε, νόσο των φυτών του οποίου στο Αφγανιστάν, αλλά μπορεί να οφείλεται και ε, κάποιες επιχειρήσεις που έγιναν με τις τουρκικές αρχές για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών αλλά είχαμε και άλλες χώρες όπως η Ελβετία, όπως συνέβη αυτό και στη Ρωσία πριν να το σχάρι όπου για να απαντηθεί αυτή η έλλειψη ηρωίνης υπάρχει μια άλλη ουσία η που χρησιμοποιούν αντί της ηρωίνης και πρόκειται για μια ενέσιμη ουσία επίσης ε, αλλά πλήττει την υγεία και αυξάνεται πολύ περισσότερο ο κίνδυνος για HIV. Πολύ περισσότερο από ό,τι με την ηρωίνη. Τι βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την αγορά των οπιούχων. Είναι εδώ αυτό που αποκαλούμε με προφανή ισορροπία, γιατί αυτό Βλέπουμε στην Δυτική Ευρωπή και στη Βόρεια Αμερική ότι η χρήση της ηρωίνης, ε, αν δεν μειώνεται, σταθεροποιείται. Στη ΣΥΠΑ, παραδείγματος χάρη, η χρήση της ηρωίνης ε, μειώνεται και βλέπουμε να διευκρίνεται η συνταγογράφηση των ε, οπιοειδών. Και τώρα στις ΗΠΑ η κατανάλωση αυτών είναι υψηλότερη από άλλα παράνομα ναρκωτικά αλλά τι βλέπετε εδώ στο γράφημα. Οι μπάρες με το καφέ είναι η παραγωγή οποίου παγκοσμίω και οι γραμμές που βλέπετε είναι οι τιμές ε, στις ε, χώρες παραγωγής και τι βλέπουμε ότι η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες ε, τις χώρες πηγή, Μιανμάρ, Αφγανιστάν, Κολομβία και πώς γνωρίζετε όταν αυξάνεται η τιμή ε, στην, σε μια οικονομία, αυτό είναι ένδειξη ότι αυξάνεται και η ζήτηση. Πώς ε, μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε ε, αυτή την ανισορροπία. Ακόμη και αν υποτιμήσουμε την καταναλωτική αγορά παγκοσμίω, υπάρχουν αγορές που μεγεθύνονται, που δεν τις βλέπουμε και μπορεί να είναι στην Ασία και στην Αφρική, καθώς δεν έχουμε στοιχεία για τις χώρες αυτές και έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια αύξηση για τα οποία χρησιμοποιούνται εκεί αλλά δεν υπάρχει ανείχνευση, ε, γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να το δείξουμε αλλά επίσης ε, μπορεί να ε, υπάρχει αύξηση της δράσης των διοκτικών αρχών. Ε, το χάρη αυτό αντικατοπτρίζεται ίσως στις αυξανόμενες τιμές ή θα μπορούσε να σημαίνει ότι η αγορά του κατέργαστου οποίου έχει της ηρωίνης να αυξάνεται. Το 2010 είδαμε μια μεγάλη αύξηση των κατασχέσεων μορφήνης στο Πακιστάν. Όπως ε, ξέρετε, η μορφή είναι μια ουσία που παράγεται πριν την ηρωίνη και ίσως ε, αυτό να αύξησε την ε, ζήτηση που είδαμε στο όπιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τιμές και πάλι, γιατί εξετάζουμε τις τιμές, γιατί οι τιμές μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα σχετικά με τις αλλαγές στην προσφορά και στη ζήτηση βλέπετε και πάλι εδώ τις μπάρες, έχουμε την παγκόσμια παραγωγή οπίου Και θα ήθελα να σας ζητήσω να προσέξετε την μπλε γραμμή. Βλέπετε στο κάτω μέρος την τιμή του οποίου στο Αφγανιστάν, ενώ η καφέ γραμμή με τα τριγωνάκια που βλέπετε, ε, να μειώνεται λίγο και μετά να μένει σταθερή, είναι η λιανική τιμή της ηρωίνης στη Δυτική Ευρώπη. Και όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπο τη τιμή του οποίου στο Αφγανιστάν, στις ε, τιμέ τη ηρωίνη στην Ευρώπη. Γιατί και πάλι αυτό είναι μία ένδειξη ότι η τιμή και η αγορά στην Ευρώπη καθορίζεται κυρίως από τη ζήτηση παρά από την προσφορά. Και βασικά η συνεχώς μειούμενη τιμή στην Ευρώπη μας δείχνει ότι η αγορά της χρήσης των χρηστών της ηρωίνης παραμένει σταθερή. Τι μπορούμε να πούμε για την κοκαίνη. Εδώ βλέπουμε τις συνήθεις οδούς που έχουμε από τις Άνδης στην Καραϊβική και στην Ευρώπη ή από τις Άνδης στην Βενεζουέλα και στην Ευρώπη μέσω της Δυτικής Αφρικής. Μία νέα οδός που βλέπουμε είναι από τη Βραζιλία στα Βαλκάνια, στη Δυτική Ευρώπη, κατόπιν. Έχουμε λοιπόν εγκληματικά δίκτυα από τα Βαλκάνια, στη Βραζιλία, που συνεργάζονται με τους Νιγηριανούς ε, στη Βραζιλία και φέρνουν κοκαίνη μέσω της Βαλκανικής Οδού στη Δυτική Ευρώπη. Και από τη Βραζιλία επίσης Βλέπουμε μία οδό προ τη Δυτική Αφρική και πάλι από τη Δυτική Αφρική δια της οδού να φτάνει κοκκινή στην Ευρώπη και από τη Δυτική Αφρική, όταν φτάσει δηλαδή στη Δυτική Αφρική, φτάνει στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη μέσω του δικτύου της Αλκάιντα στη Βόρεια Αμερική, λέει ο Μιλήτρια χρησιμοποιείται, μάλλον δηλαδή αυτή η διακίνηση διευκολύνεται από τις τρομοκρατικές ομάδες. Βλέπουμε και μια αναδυόμενη αγορά μέσω της Αργεντινής, να περνά από την Αργεντινή και δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες ε, σε σχέση με τις διεθνείς εγκληματικές ομάδες. Ε, βλέπουμε εδώ μετακίνηση από την Αργεντινή προς την ακτή της Βραζιλίας και κατόπιν φτάνουν στην Ευρώπη. Και απευθείας επίσης από τη Βραζιλία ένα αερίος προς την Ευρώπη και από την Ευρώπη έχουμε ε, έκσταση να στέλνεται πίσω. Έχουμε αυτή την ανταλλαγή κοκαίνης έκσταση. Και μια, βλέπουμε αύξηση των αποστολών κοκαίνης μέσω λιμανιών. Και επίσης έχουμε τώρα ε, διακίνηση κοκαίνης και μέσω της ε, Βαλτικής. Ε, Υπάρχουν ε, πολλά εμπορικηματοκιβώτια που στέλνονται από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν οι εγκληματικέ οργανώσει καταλάβονται αυτά τα εμπορικηματοκιβώτια. Και κάτι ακόμη για την κάναβη. Για να δούμε αν είναι μια αγορά σε μετάβαση Ευρώπη σε σχέση με την κάναβη. Ξέρετε ότι ε, η κάναβη έρχεται κυρίως από το Μαρόκο, κυρίως μέσω της Ισπανίας αλλά βλέπουμε εδώ πόσο σημαντικό είναι το, ότι η σημασία του Μαρόκου στην αγορά της Ευρώπης μειώνεται ελαφρώς, αλλά βλέπουμε αύξηση στην παραγωγή και πρόκειται για μια εγχώρια παραγωγή όπου και εκεί έχουμε διεθνείς εγκληματικές ομάδες να εμπλέκονται στην καλλιέργεια κάναβης στην Ευρώπη. Και πάλι όταν υπάρχουν κατασχέσεις, βλέπουμε ομάδες ε, που διακινούν όχι μόνο κάναβη αλλά και ροήνη και κοκαίνη. Και αυτή είναι μια ένδειξη ότι οι χώρες στην Ευρώπη που αναφέρουν αύξηση 1100 ε, ε, στην κάναβη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια πολύ γρήγορη αλλαγή στην Ευρώπη στον τομέα αυτό με εγχώρια παραγωγή. Έχω και άλλα λεπτομερή στοιχεία, αλλά νομίζω τέλειωσαν τα 15 μου λεπτά. Σα σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που απαντήσατε βάθο βάθος στο ε, θέμα αυτό και που σεβαστήκατε και τα 15 λεπτά. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρόσμπαχ που εκπροσωπεί την Ιντερπόλ που όπως σας είπα πριν θα παρουσίασει μια καθολική αξιολόγηση της οργάνωσής του σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και τις σχετικές απειλές. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ονομάζομαι Μπέρντ Ρόσπαχ και είμαι διευθυντή τη μονάδα Ειδικού εγκλήματο και ανάλυση στην Ιντερπόλ στη Λιόν, την Γαλλία. Βρίσκομαι εδώ γιατί ακριβώς οι αρμοδιότητες μου εμπίπτουν απόλυτα στον τίτλο της Επιτροπής αυτής, που πρόκειται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της νομοποίησης του παράνομου χρήματος. Καλύπτουμε επίσης και άλλους τομείς εγκλήματος, ποικίλου. Πρόκειται για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, για στιμένου αγώνες, δημόσια ασφάλεια, εγκλήματα κατά του περιβάλλοντο, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, πειρατεία στη θάλασσα, εκλοπή έργων πλαστά αγαθά, διαβατήρια, παραχάραξη χρήματο. Βέβαια, πολλοί από εσά δεν είσαστε εξοικειωμένοι με την οργάνωσή μα. Όμω πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε 190 χώρε μέλη σήμερα. Η Γενική μα Γραμματεία βρίσκεται στη Λιόν της Γαλλίας και έχουμε γραφεία σύνδεση στι Βρυξέλλες, στη Νέα Υόρκη, τον Μπένος την Πανκόκ, το Σαν Σαλβαδόρ, το Αμπιτζάν, τη Γιαουντέ, το Χαράρε και το Ναϊρόμπι. Επίσης ετοιμάζουμε μια νέα δομή στη Σιγκαπούρη όπου θα εδρεύει το Global Complex της Interpol και που πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί το 2014. Γενικό μα γραμματέα είναι ο κύριο Ρόναλτ Κανόμπλε, ο οποίο είναι από τι ΗΠΑ και πρόεδρο τη Ιντερπόλ είναι ο κύριο Ζουμπόν Χαουκού, που είναι από τη Σιγκαπούρη. Τώρα, κάθε χώρα μέλο εκπροσωπείται σε εθνικό επίπεδο. Κάθε λοιπόν ε, γραφείο μας εκπροσωπείται από άτομα από κάθε χώρα μέλος βάσει του εθνικού νόμου. Και έτσι υπάρχει 24 ώρες 24 ώρες 7 ώρες τη βδομάδα επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των εθνικών γραφείων ανά το κόσμο, αλλά και με τη Γενική Γραμματεία και όλα τα γραφεία μας όπως είπα νωρίτερα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μεταφέρουμε και να επικοινωνήσουμε μεταξύ άλλων δακτυλικά αποτυπώματα, εικόνες, προφίλ DNA κλπ. Έχουμε τράπεζα δεδομένων την οποία μπορούν να συμβουλευτούν τα μέλη μας οποιαδήποτε στιγμή. Οποιοςδήποτε χρειάζεται ε, κάποια πληροφορία από τα διάφορα εθνικά μας γραφεία για ταυτότητες ή για πυροβόλα όπλα ή για οτιδήποτε άλλο ύποπτο μπορεί να συμβουλευτεί την τράπεζα αυτή δεδομένων μας. Η Γενική μας Γραμματεία επίσης λειτουργεί 24 ώρες τώρα 7 μέρες τη βδομάδα στη Λιόν, στο Πενοσάιρες και σύντομα στην Σιγκαπούρη και μπορεί να απαντήσει σε μηνύματα και σε αιτήσει που έρχονται από τα μέλη μας στις τέσσερις επίσημες γλώσσες μας, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και ισπανικά είναι σημαντικό να ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε ένα αυτόνομο ερευνητικό γραφείο ή ανακριτικό γραφείο που μπορεί να συλλάβει ή να βάλει στη φυλακή κάποιον. Εμείς είμαστε ένα δίκτυο αστυνομίας που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο και που συγκεντρώνει ε, δεδομένα σχετικά με το διεθνές έγκλημα που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει βέβαια διάφορα εργαλεία και διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέλη μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε γενικά το οργανωμένο έγκλημα σε όλες του τις μορφές, αλλά ασχολούμαστε με διάφορες δραστηριότητες που απασχολούν τη μία χώρα και την άλλη, γιατί ακριβώ πρόκειται για διεθνές έγκλημα. Είναι μια καθημερινή πρόκληση για μας. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι χώρες μέλη να μας ενημερώνουν για τις υποψίες που έχουν ή για εγκληματικές ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους από ένα περισσότερο άτομα. Πρόκειται δηλαδή για καθημερινή ανταλλαγή απόψεων που έχουμε με τις χώρες μέλη. Για ορισμένους τομείς εγκλημάτων φαίνεται ότι το οργαμένο έγκλημα απαιτεί ειδικέ στρατηγικές από κοινού μεταξύ ημών και των μελών μας. Βάζουμε βέβαια προτεραιότητες σε διάφορους τομείς εγκλήματος και εκεί αυτούς τους τομείς τους αναθέτουμε στο προσωπικό μας, άλλοτε με βραχυπρόθεσμες και άλλο με μακροπρόθεσμες ενέργειες και προγράμματα. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά μια που είμαστε διεθνής αστυνομία, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις στη δημόσια ασφάλεια και στο κράτος ε, δικαίου από μόνοι μα. Γι' αυτό ακριβώς συνεργαζόμαστε και έχουμε συμφωνίες ε, συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς, είτε με την UNODOC, την οποία μόλις ακούσατε, με τη Διεθνή Οργάνωση Τελωνίων, με την, τον ΠΟΕ, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και με διάφορες περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Europol, η ΣΕΠΚΑ, που αφορά την νοτιοανατολική Ευρώπη και την αστυνομία της, το ΚΑΡΕΚ, που αφορά τις μυστικές υπηρεσίες της Ασίας και άλλες οργανώσεις αστυνομίας. Σε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχέσεις μας δεν είναι απλώς ανταλλαγή επιστολών ή μνημόνια κατανόησης. Στην πραγματικότητα πηγαίνουμε ακόμα πιο μακριά και έχουμε σε πραγματικό χρόνο συνεργασίας ε, για θέματα αστυνομικής έρευνας. Δυστυχώς βέβαια δεν έχω αρκετό χρόνο εδώ για να σας αναφέρω όλους τους τομείς εγκλήματος που καλύπτει η Ιντερπόλ και αυτό προτείνω να αναφερθώ μόνο στα, στους κύριους τομείς που ενδιαφέρουν εσάς. Όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εκτενείς δραστηριότητε μας, σας συστήνω να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, η οποία καθημερινά ενημερώνεται. Όσον αφορά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τα παράνομα ναρκωτικά. Εμείς ασχολούμαστε με την παραγωγή και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, κυρίως σε χώρες όπως το Μεξικό, όπου υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη βία και διαφθορά η κυβέρνηση προσπαθεί βέβαια να τα αντιμετωπίσει, αλλά έχει τεράστιες προκλήσεις μπροστά της όσον αφορά και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και είναι κάτι που αφορά όχι μόνο το Μεξικό, αλλά και άλλες περιοχές όπως είναι η Νοτιοανατολική Ασία. Διάφορες ε, πάντως εγκληματικές οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να επιβάλλουν το δικό τους νόμο. Στην Ευρώπη επίσης καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα το λαθρεμπόριο ηρωίνη κυρίω που προέρχεται από το Αφγανιστάν. Η εταίροι μας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αυτού είναι οργανώσει που σας ανέφερα πριν. Επίσης έχουμε ειδικέ σχέσεις με χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Γαλλία, στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, του Παρισιού. Για την Αφρική επίσης η Ιντερπόλ δραστηριοποιείται και εκεί όσον αφορά την ε, κοκαίνη που περνάει από εκεί και που προέρχεται από την ε, Νότια Αμερική και καταλήγει στην Ευρώπη. Έχουμε διαπιστώσει επίσης ότι η παράνομη παραγωγή μεθαμφεταμίνης αυξάνεται πάρα πολύ τελευταία. Έχει φτάσει σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και περνάει από την Αφρική, το Ιράν και την Ανατολική Ασία. Το οργανωμένο έγκλημα τώρα στην Ευρώπη δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς που καταπολεμούμε εμπορία ανθρώπων για παράδειγμα, κλοπή ε, κοσμημάτων, ε, κλοπή έργων τέχνης και πολλά άλλα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα προγραμμάτων που εμείς έχουμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται όρος Πάνθυρας και ο οποίος ε, αντιμετωπίζει την κλοπή υψηλής αξίας κοσμημάτων στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή αλλά και σε ορισμένες σχετικές χώρες. Τα αυτά ε, λαμβάνουν χώρα από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που έχουν τη βάση τους κυρίως στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρατηρούμε λοιπόν τις δραστηριότητές τους και διαπιστώνουμε ότι επεκτείνουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες πέρα από την περιοχή όπου αρχικά εντοπίστηκαν. Και αυτό το έχει διαπιστώσει η Interpol παρακολουθώντας από την αρχή με το πρόγραμμα αυτό. Επίσης έχουμε το πρόγραμμα Millennium, το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει ε, διασυνοριακά εγκλήματα από την Ευρώπη και την Ασία κυρίως. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα στον τομέα αυτό και δεν πρόκειται μόνο για τη συλλογή πληροφοριών εδώ. Πιο πρόσφατα η Ιντερπολ και η ομάδα της, η Ερμόδια για αυτό, το 2012 αναπτύχθηκε στη Λιμός της Γαλλίας για να βοηθήσει την γαλλική αστυνομία και την Europol σε μια δράση που ονομάζεται δράση κόσμημα, που είχε σαν στόχο εγκληματικέ ομάδε από τη Γεωργία και την Αρμενία και συνελήφθησαν 21 άτομα. Υπάρχει επίση και το πρόγραμμα BESA, το οποίο συμπλήρωσε τη διετή εντολή του και ασχολήθηκε κυρίω με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ιντερπόλ συνεργάζεται στενά με τι οργανώσει που σα ανέφερα πριν, τη ΕΠΚΑ για παράδειγμα, σε επίπεδο ανάκριση αλλά και επιχειρησιακό αλλά και μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε κάθε χρόνο αποτελέσματα τα οποία αναλύει η Ιντερπόλ υπό την μορφή ειδικών αξιολογήσεων που ονομάζονται ΣΕΤΑΚ. Οι αναλύσεις αυτές φτάνουν και στην ΣΕΠΚΑ και εντοπίζουν τα θετικά και τις αδυναμίες μέσα βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούμε. Περιτώ να πω ότι οι εκθέσεις ε, αυτές είναι χρήση της αστυνομίας μόνο. Επίσης, ε, έχουμε και την εμπορία ανθρώπων. Και εδώ έχουμε πολλές εγκληματικές οργανώσεις που ασχολούνται σε αυτό και που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την δραστηριότητα. Τα θύματα τα βρίσκουν κυρίως σε χώρες που έχουν ιδιαίτερα δύναμες οικονομίες και όπου υπάρχει πολιτική αστάθεια και πολλές φορές ε, και ε, διενέξεις και σειράξεις. Το θέμα της εμπορίας ε, ανθρώπων μας απασχολεί όλος ιδιαίτερος γιατί εμπλέκονται και παιδιά εδώ. Παιδιά τα οποία χρησιμοποιούνται για διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Συνεργαζόμαστε επίσης με διάφορες περιφερειακές οργανώσεις και σε αυτό το τομέα. Συνεργαζόμαστε για παράδειγμα με τη Frontex. Η Interpol επίσης δραστηριοποιείται για να αντιμετωπίσει και το οργανωμένο έγκλημα όσον αφορά τα στιγμένα παιχνίδια και τα παράνομα στοιχήματα που γίνονται για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Υπάρχει μια ειδική ομάδα η οποία ασχολείται με τον συντονισμό ε, της έρευνας στον τομέα αυτό. Έχουμε επίσης και το λαθρεμπόριο πλαστών ε, προϊόντων και παράνομων φαρμάκων. Και αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα για την Ιντερπόλ που έχει μια ειδική ομάδα για τα φαρμακευτικά προϊόντα και προσπαθεί να συντονίσει τις ε, δράσεις για την καταπολέμηση αυτής της απειλής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είμαστε αποτελεσματικοί. Είχαμε τελευταία μία ε, δραστηριότητα, μια δράση μάλλον, την οποία ονομάσαμε Παγκαία, η οποία μέσα σε μία εβδομάδα συντόνισε τις δράσεις σε 80 χώρες μέλες και κατέληξε να κλείσει 13.500 ιστοσελίδες, να κάνει κατάσχεση 8.000 ε, ε, πακέτων που περίχανε πλαστά ή παράνομα φάρμακα και κατήσχε επίσης και 2,4 εκατομμύρια δόσεις παράνομων φαρμάκων από 48 χώρες. Η Ιντερπόλ αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τα δίκτυα μεταφοράς των λαθρεμπόρων ατόμων, για παράδειγμα. Και έτσι προχωρούν στις τρομοκρατικές τους δραστηριότητες, οι οποίες βέβαια απειλούν την δημόσια ασφάλεια στις χώρες μας. Έχουμε μια ε, κοινή πρωτοβουλία που αναλάβαμε πρόσφατα για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Και ενθαρρύνουμε 190 χώρες μέλη μας να καταρτήσουν ειδικέ μονάδες που να χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό και που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ιντερπόλ, σε συνεργασία δηλαδή με την Interpol, να προχωρήσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα δίκτυα. Όπω είπα και πριν, είναι μια καθημερινή πρόκληση για μα για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα διεθνώ. Η Interpol αγωνίζεται για να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή με του τεχνικού αλλά και του ανθρώπινου πόρου που διαθέτει, έχει αναπτύξει ίδια. Βέβαια, δεν έχουμε όλοι τα ίδια μέσα. Παρ' όλα αυτά, Ό,τι εμπόδια και αν υπάρχουν μπροστά μα δεν μας σταματάνε. Στην πραγματικότητα η διεύθεσή μα στατικικού σχεδιασμού δουλεύει καθημερινά για την ε, ανάπτυξη των κατάλληλων συνθήκων ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας βρίσκοντας τις κατάλληλες λύσεις είτε πρόκειται για συλλογή δεδομένων είτε για δράσεις. Επίσης προσπαθούμε να έχουμε και πόρους οι οποίοι να πηγαίνουν κατευθείαν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το εύκολο και το γρήγορο κέρδος από παράνομες δραστηριότητες. Η εθνική νομοθεσία όμως πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα και να υπάρχουν όμως και κατάλληλοι πόροι για να αντιμετωπιστούν. Μόνο μέσω μιας συντονισμένης δράσης σε συνεργασία με την Europol, την UNODOC και άλλες οργανώσεις θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρόσμπαχ. Τελειώσατε και ένα λεπτό νωρίτερα. Όπως είχα, έχω ήδη λοιπόν πει, τώρα θα έχουμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ε, μπορούν να ερωτήσουν οι συγητές ε, και οι συντονιστές. Ε, θα απαντήσουν οι ομιλητές και εάν τα καταφέρουμε θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα είμαι σίγουρα μέσα στα δύο λεπτά που μου διαθέσατε. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ε, δύο εισηγήσεις. Άκουσα όλα αυτά τα οποία ε, παρουσιάστηκαν στις παρεμβάσεις τους και, και από τα δύο λοιπόν και από τις δύο εισηγήσεις προέκυψε ένας κοινός παρονομαστής η σχέση μεταξύ την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία η Αλκάιντα ε, έχει άμεση σχέση με, την, ε, με τα ναρκωτικά και με την με πώληση ναρκωτικών. Αναφέρθηκε αυτό στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη αναφέρθηκε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να αντιμετωπιστούν και τα δύο αυτά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν τίθεται σαφώς το εξής ερώτημα, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είναι απολύτως σαφές και το ανέφερα. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς που είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν και το οργανωμένο έγκλημα και τον, ε, την τρομοκρατία στις ε, διάφορες εκφάνσεις της. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα όρια. Υπάρχουν όρια συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, ε συμφωνίες για, τον, για την τρομοκρατία. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν, χάρη μεταξύ άλλων το SWIFT. Και ποιες είναι οι ενδείξεις που υπάρχουν έτσι ώστε να μην εμφανίζονται όρια στη συνεργασία ανάμεσα στις ε, αστυνομικές αρχές που είναι οι πρωταγωνιστές για να αντιμετωπίσουν ε, το εγκληματικό αυτό φαινόμενο και για να μπορούν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά προς την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών. Γιατί οι διαδρομές τους αλλάζουν ε, σύρεχώς, όπως και οι ε, διαδρομές ε, των ε, οργανωμένων κλιματιών που φτάνουν στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό από την Νότια Ευρώπη. Μποργκέτσιο, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει μια τρέχουσα επικαιρότητα και αυτή μας καλεί να εξετάσουμε μια πολύ σημαντική πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος. Αναφέρομαι στις ε, παράνομες οργανώσεις. Αναφέρομαι κυρίως σε πολύ σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα και έχουν σχέση με ε, μεταφορά ε, μεταναστών, παράνομων μεταναστών μέσα από πολύ επικίνδυνους ε, δρόμους. Ένα λοιπόν κομβικό στοιχείο για να αντιμετωπίσουμε την μετακίνηση των παράνομων μεταναστών είναι να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τα οικονομικά συμφέροντα που οδηγούν ε, σε αυτές τις μετακινήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, την εκπρόσωπο της Ίντερπολ. Ποιες είναι οι στρατηγικές της Ίντερπολ για να εντοπίζονται οι οργανώσεις αυτές, όπως και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν και που επιτρέπουν στις ε, εγκληματικές οργανώσεις να εκμεταλλεύονται αυτό το φαινόμενο που είναι ένα από τα πραγματικά πλέον απάνθρωπα που μαστίζουν σήμερα την ανθρωπότητα. Για δύο λεπτά ο κύριος Ματιέ. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τους δύο μιλητές ε, για την πλήρη παρουσίασή τους ε, και για τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας του οργανωμένου κλίματος ε, και της διακίνησης ναρκωτικών. Κυρία Μέ, Καταρχήν να σας θέσω μια ερώτηση. Ξέρω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναλάβει να καταπολεμήσουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να μου πείτε Ποια είναι η βοήθεια που προσφέρει ο οργανισμός στα κρατημέλη, ε, σε ποιο συχνή βάση πρόκειται για νομική βοήθεια, πρόκειται για μια βοήθεια που αφορά περισσότερο όχι την επιχειρησιακή καταπολέμηση αλλά επιτόπου και θα ήθελα να μου πείτε τι, τι, τι ζητούν περισσότερο τα κρατη από εσά και επίσης ε, ξέρω ότι υπάρχει μια απόσταση ε, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια διευκρίνηση για το θέμα αυτό και επίσης ε, ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα ε, υπάρχει σύνδεση πολιτικής σταθερότητας με την κατανάλωση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης είδατε σαφή μείωση, μία ρήξη σε ό,τι αφορά την κατανάλωση των ναρκωτικών και κύριε Ρόσμπακ από την Ιντερπολ. Θα θέλα να μας πείτε λίγο περισσότερα για τα συνθετικά ναρκωτικά. Έχετε κι εσείς μια ξεκάθαρη αποστολή για την καταπολέμηση ε, των εργαστηρίων που παρασκευάζουν αυτά τα συνθετικά ναρκωτικά. Θα ήθελα να μας ε, πείτε δύο λόγια για το πώς συνεργάζεστε με την Europol πώς ε, εργάζεστε με την Europol και με την Eurojust σε τι συνίσταται η συνεργασία σας και ε, εσείς αντιμετωπίζετε όπως και η Europol ε, δυσκολία στην εξέβρεση πληροφοριών που πρέπει να σας δίνουν τα κράτη-μέλη γιατί εργάζεστε κατά κάποιο τρόπο ε, σε έναν κόσμο απορρίτου. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές οι ανταλλαγές πληροφοριών μπορεί να είναι κάπως πολύπλοκες μεταξύ ορισμών κρατών όλων και του δικού σας οργανισμού. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν από αυτού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα λοιπόν, ε, εκ μέρους της ε, Γκουε, Σόντεγκαρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω λοιπόν μία ερώτηση προς την κυρία Με. Θα ήθελα να γνωρίζω Ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, από την εισβολή στο Αφγανιστάν μετά το 2001. Αυξήθηκε η παραγωγή επειδή υπήρχαν ίσως ε, περισσότερα χρήματα ή μειώθηκε η παραγωγή ή δεν υπήρξε καμία απολύτως επίπτωση. Και η δεύτερη ερώτησή μου προς τον κύριο Ρόσμπαχ πρόκειται εδώ για δύο θέματα που έχουν σχέση με την ε, ερώτηση σχετικά με την Europol. Υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία με την Europol και αν υπάρχουν, ποια είναι αυτά, θα θέλαμε να ενημερωθούμε. Ξέρω ότι οι δύο φορείς ε, συνεργάζονται με αγαστό τρόπο, ε, αλλά μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα ήθελα να γνωρίζω. Άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με το ξέπλυμα του χρήματος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο οργανωμένο έγκλημα. Το θέμα δεν είναι μόνο να εισπράξει κανείς ε, το παράνομο χρήμα, αλλά και να το νομιμοποιήσει, να το ξεπλύνει όπως λέμε. Κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είδαμε ότι καθόλου αξιοπρεπείς εταιρείες και τράπεζες δέχονται να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Κύριε Κόπ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να πω ότι ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις, όχι μόνο γιατί παρέμειναν μέσα στο χρόνο που τους είχε δοθεί, αλλά και γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω μία ερώτηση ε, και προς τους ε, δύο ομιλητές. Έχει σχέση με την ε, πολιτική δίωξη οργανωμένων κλίματος ναρκωτικών. Και Ερωτώ, όσον αφορά τον εντοπισμό διακίνησης ναρκωτικών, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εντοπιστούν τα ναρκωτικά αυτά ε, μέσα από πληροφορίες ή ε, συστήματα που έχουν σχέση με το PNR, ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις διοκτικές αρχές. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εντοπιστεί το θέμα αυτό. Και κάτι άλλο. Ε, νομίζω η πρώτη ομιλήτρια αναφέρθηκε στην τιμή των ναρκωτικών. Κόστος ε, και τιμή, σχέση κόστους τιμής και ρωτώ, κατά την άποψή της υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στις ε, πολιτικές ε, που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση των ναρκωτικών και την απόκτηση ναρκωτικών. Υπάρχει λοιπόν σχέση αυτών με το κόστος και με το όφελος μπορεί να έχει κανείς ε, προμητεύοντα αγορές με αυτά τα ναρκωτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους των Πρασίνων. Στάσε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να Ευχαριστώ του μελητές για όλα αυτά που μας είπαν. Ε, να αναφερθώ στη συνεργασία των θεσμών. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Εξάλλου, θα ήθελα να ενημερωθώ και, και για κάτι άλλο που με απασχολεί. Αφορά την Ίντερπολ κυρίως. Εσείς πώς ακριβώς καθορίζετε τις ε, μεθόδους εργασίας σας. Πώς ακριβώς ασκείτε το δημοκρατικό έλεγχο. Δεν είναι ότι αμφισβητώ τις ε, καλές σας προθέσεις, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά τις ε, έρευνες θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ελέγχου και επαλήθευσης και ε, κυρίως επειδή εσείς εκπροσωπείτε έναν οργανισμό που δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι άλλοι. Ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνομαι στην κυρία εκ μέρου των Ηνωμένων Εθνών. Μιλήσατε στην αρχή για το δίκτυο τη Αλκάιντα στη Βόρειο Αμερική. Μήπω εννοούσατε Βόρειο Αφρική. Κάπω πρέπει να το διευκρινίσετε. Και ε, δεύτερη ερώτηση. Κατά τη δική σας άποψη, τι πρέπει να κάνουμε που δεν κάνουμε για να λύσουμε τα προβλήματα. Τώρα, προς τον κύριο της Ιντερπολ απευθύνομαι. Δεν αναφέρατε την Κίνα, ούτε την ε, γλώσσα, την κινέζικη. Η Ιντερπολ ε, συνεργάζεται με τους ε, Κινέζους, γιατί δεν το αναφέρατε καθόλου αυτό. Άλλη ερώτηση. Εσείς, κατά τη δική σας άποψη, τι πρέπει να κάνουμε που παραλείπουμε αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μια άποψη από αυτού, όπως έχουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Και άλλη ερώτηση. Αυτά τα κέρδη τα οποία προσπορίζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πού πάνε. Σίγουρα δεν μπαίνουν μέσα στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Πέστε μας λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα, τα παράνομα, πού ακριβώς διοχετεύονται. Ευχαριστούμε τον κύριο Νιούτον Ντάν. Τώρα δύο λεπτά, Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι ε, παρακολουθώ την κατάσταση όσον αφορά αυτό που αποκαλείται drug cut. Εμείς στη Σουηδία έχουμε πρόβλημα με τους Σομαλούς. Όπως ξέρετε η οργάνωση αυτή είναι απαγορευμένη στην Ολλανδία, αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι, το Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπως μπορείτε να δουλέψετε, να μας πείτε λιγάκι κάτι από αυτού, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με την ε, κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Σουηδίας και υπάρχουν ε, σχέσεις ανάμεσα στην Al-Shabaab που διοχετεύει ε, το Λονδίνο ή το Σίπχολ του Αμστερνταμ ναρκωτικά και μετά αυτά διοχετεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα χρήματα που συγκεντρώνονται ε, διοχετεύονται πίσω στην Al-Shabaab για τρομοκρατικές ενέργειες. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας ενημερώσετε επ' αυτού. Αν έχετε παρακολουθήσει λιγάκι τις διαδρομές του χρήματος, δηλαδή τελικά από τα χρήματα που συγκεντρώνονται, ε, σε τι ακριβώς διοχετεύονται. Ε, τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας πέντε λεπτά ο καθένας ε, για να δώσουμε μετά το λόγο σε άλλους ευρωβουλευτές που έχουν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Ρόσμπαχ. Κυρία Μέτ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Ε, ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όλες. Καταρχήν, τι μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι αυτή ήταν μια καινή ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, αλλά και γενικά. Κάθε φορά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση σε μια οδό, ανακύπτει μια καινούργια. Κάθε φορά που προσπαθούμε να περιορίσουμε τη διακίνηση κάποιων ναρκωτικών, εμφανίζονται νέα ναρκωτικά. Έχουμε νέε παράνομε ουσίε κτλ. Να αναφερθώ λοιπόν σε κάποιε ερωτήσει προ την κατεύθυνση αυτή και να αναλύσω τι μπορούμε να κάνουμε. Μία σημαντική πτυχή είναι η διαφθορά. Όταν σας έδειξα όλους τους οδούς, ε, είναι δυνατές αυτή η οδή, γιατί υπάρχουν διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, οι οποίοι αφήνουν τα ναρκωτικά να περνούν από τις χώρες. Και αυτό είναι από τα κυρία στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε ε, να σταματήσουμε τη διακίνηση από τη μια χώρα στην άλλη. Ένα άλλο ζήτημα προς αντιμετώπιση είναι τα νομικά εργαλεία, τα νομικά μέσα. Υπήρξε μια ερώτηση, τι κάνουμε εμείς ε, ως Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, ε, προσφέρουμε νομική βοήθεια στις χώρες μέσω διάφορων ε, μοντέλων ή τουλάχιστον τις βοηθούμε για να διασφαλίσουμε ότι είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα νομικά μέσα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, πάντοτε αυτός είναι ο κινούμενος στόχος, γιατί όπως είπαμε και πριν, όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ναρκωτικό, έρχεται ένα άλλο ναρκωτικό και τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα νέα ναρκωτικά. Να σα χάρη το ίδιο για τι τρομοκρατικέ δραστηριότητε, Ξέρετε, αλλάζουν οι τρόποι δράση συνεχώ. Έτσι λοιπόν και το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να αλλάζει με την ίδια ταχύτητα, όπως και περάνομες δραστηριότητε. Ένα άλλο ζήτημα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω κάποιος ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη και τι συμβαίνει με όλα αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Προηγουμένω ε, δεν είχα χρόνο να σα δείξω μια διαφάνεια, αλλά θέλω να σα πω ότι ε, όταν μιλάμε για κατασχέσει ναρκωτικών, ε, αν δούμε την παραγωγή και την ποσότητα των ναρκωτικών που έχουν κατασχεθεί, βλέπουμε ότι για την ηρωίνη, παραδείγματο χάρη, έχουμε μεταξύ 20 και 30% της ηρωίνης που παράγεται να είναι υποκατάσχεση τελικά να τίθεται υποκατάσχεση. Το 20% δηλαδή αφαιρείται από την αγορά από τις διοικητικές αρχές. Για την κοκαίνη είναι ακόμη ψηλότερο το ποσοστό. Είναι μεταξύ του 30-40-50% όλης της ε, ε, κοκαίνη ε, που ουσιαστικά κατάσχεται από τις ιδιωτικές αρχές. Αν δούμε τώρα την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. ή αν θέλετε αυτά τα βρώμικα χρήματα. Μόνο 0,3-0,5% όλων των χρημάτων, όλων των κερδών που προέρχονται από τις παράνομες δραστηριότητε που κερδίζουν αυτές ε, οι εγκληματικές ομάδες ανοιχνεύεται. Έτσι λοιπόν ε, πρόκειται για τον τομέα όπου οι εγκληματίες συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Στην πηγή νομίζω πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να δούμε πώς γίνονται αυτά τα κέρδη και πώς μπορούν να ανακυκλωθούν. Γιατί, τι βλέπουμε, ότι το οργανωμένο έγκλημα τώρα ουσιαστικά έχει τις παρισφρήσεις στις νόμιμες δραστηριότητες και βλέπουμε μια οργάνωση που μπορεί να συμμετέχει σε μια παράνομη δραστηριότητα, αλλά όλα είναι και περισσότερο βλέπουμε οργανώσεις που βρίσκονται στο όριο μεταξύ νόμιμων και παράνομων δραστηριοτήτων. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να παρέμβουμε για να σταματήσουμε τη ροή των χρημάτων και των κερδών. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Νομίζω ότι υπήρξε και μια ερώτηση σχετικά με την πολιτική περί ναρκωτικών. Αν κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει τα κέρδη των ε, παράνομων οργανώσεων. Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν ε, εξαιρετικό ταλέντο στο να αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα το modus αλλά και το τομείς που βλέπουν δυνατότητες. Δηλαδή, αν ε, σήμερα ε, είναι ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό, αύριο θα βρουν άλλο ναρκωτικό που να αποφέρει κέρδη ή μια άλλη παράνομη δραστηριότητα. Τα παράνομα στοιχήματα, παραδείγματο χάρη, τον τζόγο. Αναφέρομαι ότι το οργανωμένο έγκλημα μπαίνει σίγουρα σε αυτό το τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν ε, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και μια διμερή συζήτηση για να πέντε στις ερωτήσεις, ε, γιατί δεν πρόλαβα. Ναι, θα υπάρχει και ένας δεύτερος γύρος. για τις ε, ερωτήσεις, ίσως θα μπορέσετε να συμπληρώσετε. Ο κύριος Ρόσμπαχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, αυτό που είπατε σχετικά με την εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος με την ε, τρομοκρατία. Ισχύει το εξής, εμείς ε, ως Interpol ε, έχουμε πρόβλημα να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και νομίζω το είπα και στην ομιλία μου. τα κράτη-μέλη πράγματι αντιμετωπίζουν διαφορετικά το οργανωμένο έγκλημα. Πολλά εξ αυτών δεν είναι σε θέση να μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ακόμα και για απλά θέματα, όπως είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα ή χαρακτηριστικά των υπόπτων, για να μπορούμε τα στοιχεία αυτά να τα αποθηκεύσουμε στις τράπεζες δομένων και ενδεχομένως να τα ανακαλέσουμε. Σημασία έχει και ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, άλλο θέμα πάλι το, η τρομοκρατία. Για την τρομοκρατία υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες μονάδες όπου όμως η συνεργασία δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη γιατί όσο μεγαλύτερος ο κύκλος ε, των ε, ατόμων που γνωρίζουν πληροφορίες τόσο λιγότερες πληροφορίες δίδονται. Αυτό λοιπόν ως Interpol ε, το έχουμε δυστυχώς κατά νου. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του δημοκρατικού ελέγχου. Σε μας λοιπόν ισχύει το εξής. Εμείς εκπροσωπούμε τα κράτη-μέλη τα οποία κρατημέλη έχουν τα ε, κεντρικά τους γραφεία, εκπροσωπούνται με τους επικεφαλείς των κεντρικών γραφείων και προφανώς με τον τρόπο αυτό ε, αναλαμβάνουν άμεσα την ευθύνη. Μετά υπάρχουν ε, και άλλα όργανα όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Υπάρχει η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μια φορά το χρόνο και ε, στηρίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή με ερετούς ε, μετέχοντες επιπρόσθετα. Έχουμε και μια ανεξάρτητη επιτροπή που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες. Αυτή λοιπόν εξετάζει το θέμα και κάτω από το πρίσμα της ε, προστασίας ε, δεδομένων και σε αυτήν απευθυνόμαστε οποτεδήποτε χρειαζόμαστε νέα στοιχεία. Επειδή λοιπόν αναφέρομαι στη συνεργασία, να πω και το εξής. Αναφέρθηκε προηγουμένως η Κίνα. Βεβαίως και η Κίνα είναι ένα πολύ σημαντικό κράτος μέλος της Interpol. Νομίζω ότι το υπενήχθη αυτό, εκεί που μίλησα για το οργανωμένο έγκλημα γιατί έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τις ε, ασιατικές αρχές. Και μέσα λοιπόν από αυτές τις ε, επαφές ε, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και εμείς τη δική μας υπεραξία στις έρευνες που γίνονται στην Ευρώπη, κυρίως για τα στημένα παιχνίδια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ισορροπημένη συνεργασία ε, και πολλά απόρριτα στοιχεία σε πάρα πολλές αθλητικές εκδηλώσεις συνεργαζόμαστε στενά για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως, τα στημένα παιχνίδια. Ε, όσον αφορά τώρα την Ευρώπη. Ή έχουμε την Ευρωπόλ, την Eurojust αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας είπα ότι όλοι αυτοί οι φορείς είναι πολύ σημαντικοί για μας. Υπάρχει συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Europol και την Interpol. Εν τω μεταξύ η συνεργασία έχει ενισχυθεί περαιτέρω και με αυτά τα δύο άτομα που αναφέρθηκαν τα ονόματά τους ε, προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν τομείς που τους έχουμε εντοπίσει από κοινού. Ε, χάρη, στο κυβερνοέγκλημα, εκεί υπάρχει άμεση συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών και προσπαθούμε να επιτύχουμε το μέγιστο. Τώρα, αν ε, με ρωτάγατε για τα μειονεκτήματα, πράγματι πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχουν δυσκολίες ε, που έχουν κυρίως σχέση με την επεξεργασία των πληροφοριών. Γιατί ακόμα και αν γίνει αποδεκτό εμείς η Interpol να είμαστε εταίρος σε ένα οργανωμένο στην έρευνα για το οργανωμένο έγκλημα, εμφανίζονται τα κράτη-μέλη ε, τα οποία πρέπει να πιστούν να μας δεχτούν. Τώρα, όσον αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά, υπάρχει μια ειδική ομάδα εργασία που ασχολείται με αυτό το θέμα και ως ε, εκ τούτου έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, διεθνούς συνεργασίας ε, και με τα Ηνωμένα Έθνη. Μπορούμε και να οργανώσουμε και ακροάσεις και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων. Έχω κατά νου το χρόνο και γι' αυτό θέλω να κάνω μόνο άλλη μία παρατήρηση. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος. Πράγματι, εδώ ερχόμεθα αντιμέτωποι με μία σημαντική πρόκληση. Και υπάρχουν πολλές δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά ε, για να είμαστε Αποτελεσματική πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και τις δικαστικές αρχές. Δυστυχώς μερικές φορές ε, υπάρχουν παράλληλες έρευνες, ας πούμε, περίπτωση Μπενάλη για την Τινησία. Η Ιντερπολ ε, θα μπορούσε να εμφανίζεται ε, σε ουδέτερο έδαφος και το έκανε εκπροσωπώντας τα κράτη-μέλη. Πάμε λοιπόν σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων και δίνω το λόγο στον κύριο Ντεγιάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για την κυρία Μέα από το UNDC. Στο παρελθόν, όταν εργάστηκα για την Ολλανδική κυβέρνηση, πέρασα πολλέ εβδομάδε στη Βιέννη και μπορώ να σα πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το έργο του UNDC. Όμω, ε, στον τομέα των ναρκωτικών ε, πάντοτε είχαμε πρόβλημα, ξέρετε, ως ε, κατοχώρες, ε, δηλαδή δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τα ΗΕ μεταξύ της κάναβης και των σκληρών ναρκωτικών, όμως πρόσφατες από πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής έγιναν δηλώσεις ότι θέλουν να έχουν μια διαφορετική πολιτική για τα μαλακά ναρκωτικά και αν ε, λάβετε ε, υπόψη μια προσέγγιση κόστους αποτελέσματος ε, πράγματι δεν αξίζει να έχουμε τόσους πόρους και να κάνουμε τόσο κόπο για να καταπολεμήσουμε τα μαλακά Έχετε κάποιες μελέτες ήδη ε, στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών που να περιλαμβάνουν αυτή την ιδέα. Και σε ό,τι αφορά την νομοποίηση παράνομων εισόδων, άκουσα την απάντησή σα, αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτή την επιτροπή εδώ είναι πολύ συγκεκριμένε προτάσει σχετικά με το ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε εδώ στην Ευρώπη. Γιατί τόσο είπατε είναι κάπω γενικά. Δηλαδή, πράγματι βλέπουμε επέκταση στην οικονομία και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να αναλάβουμε για να μπορέσει και η Ευρώπη να είναι πραγματικό εταίρος του Αιγαιών Ευχαριστώ. Δύο λεπτά στον κύριο Αντίτσεβιτς. Στην κυρία Αντίτσεβιτς, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι η υπεκοσμιοποίηση αποτελεί και ευκαιρία αλλά και πρόκληση για αυτές τις παραδοσιακές ομάδες ε, του οργανωμένου εγκλήματος και ίσως ε, οι εγκληματικές ευκαιρίες σήμερα να βρίσκονται σε τομείς όπου δεν υπάρχει επαρκής ρύθμιση ε, το να πούμε ότι οι ίδιες οι ομάδες έχουν γίνει λιγότερο σημαντικές ε, από τις αγορές ε, στις οποίες δραστηριοποιούνται, ίσως είναι κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε. Φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα να κάνουν το άλμα από το να επικεντρωθούμε στις ομάδες, το να επικεντρωθούμε στις αγορές η δράση του οργανωμένου κλίματος θεωρείται ω δραστηριότητα κάποιων ατόμων παρά ω μια αγορά που έχει το δικό τη δυναμισμό. Η διαφθορά υψηλού επίπεδου συχνά υπάρχει και είναι αυτό ένα απόλυτα σαφέ. Ε, το κύριο αντικείμενο στο είναι η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών όμως καθίσταται δύσκολη η ανταλλαγή των πληροφοριών, όμως αυτό σημαίνει ότι πολλές χώρες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις ε, στον χώρο του εγκλήματος. Και τα χρήματα που μπορούν να μετακινήσουν αυτές οι ομάδες με πολύ εύκολο τρόπο μέσω του τραπεζικού συστήματος, ε, καθιστούν ε, δύσκολη την ανείχνευση αυτών των συναλλαγών. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι κάποιες τράπεζες είναι πλυντήρια για αυτά τα χρήματα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, γιατί η κατάσταση έχει όχι εξή. Η ευρωπαϊκή κοινότητα, η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει να συνεχίζεται πλέον η κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορσελίνο για δύο λεπτά. Να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη σαφήνεια των παρουσιασεών σας. Μια ερώτηση θέλω να θέσω και στους δύο μιλητές. Έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, και για τη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος, ε, αυτοί τρέχουν ε, μπροστά και εμείς ε, από πίσω. Αναρωτιέμαι τι γίνεται σε επίπεδο πρόληψης, γιατί θα ήταν πολύ πιο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό να δώσουμε προσοχή και στην πρόληψη, δηλαδή πώς θα προλάβουμε τι κάνουν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει, γνωρίζουμε τις οδούς, αλλά τις καταγράφουμε. Γνωρίζουμε τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά πώς ε, θα τις ε, καταγράψουμε. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να φερθώ σε ένα γεγονό που έγινε στη Σικελία πριν κάποια χρόνια, στη διακίνηση και στη χρήση των ναρκωτικών, ε, αλλά στο να υπάρχει προσωρινή καταπολέμηση, αν θέλετε, του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, σε αυτό ε, συνεισφέρε όταν ε, ανοιχνεύτηκε το εργαστήριο στο Παλέρμο και υπήρξε μια δουλειά μυστικών υπηρεσιών εκεί για να βρεθεί αυτό το εργαστήριο που παραγόταν ηρωίνη και κοκαίνη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτό. Και θα ήθελα να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κανόνες ε, για τη χρήση των ναρκωτικών. Υπάρχει μια ανάλυση, κάποια στατιστικά στοιχεία που να μας λένε τι λειτουργεί καλύτερα, αν είναι η απελευθέρωση ή η απαγόρευση των ναρκωτικών. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Μακλάριν δύο λεπτά. Μακλάρκιν δύο λεπτά. Um, Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, οι παραδοσιακές μέθοδοι του οργανωμένου εγκλήματος ε, σε σχέση με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που χρησιμοποιείται τώρα για να νομιμοποιούν το παράνομο χρήμα. Έχει αλλάξει δηλαδή η μέθοδος που χρησιμοποιούν εσείς, έχετε αλλάξει τις δικές σας τις ε, μεθόδους ανάλογα. Τι κάνετε για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που είναι ένας, μια νέα μορφή δραστηριότητάς τους. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μακλάρκιν. Δύο λεπτά ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλές ε, ερωτήσεις ε, τέθηκαν ε, ιδίως προς την εκπρόσωπο του Γιάννου για το ρόλο των τραπεζών. Εγώ θα ήθελα απλώ ε, να επιστήσω την προσοχή σας σε πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις του τελευταίου διευθυντή του κυρίου Αντώνιο Κώστα για αυτό το ζήτημα που είναι τόσο ευαίσθητο. Ο κύριος Κώστα είπε ρητός, εμείς έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία, έχουμε τις αποδείξεις ότι οι τράπεζες συγκεκριμένα έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μας είπε ο κ. Κώστα ότι ενεργός ο ρόλος αυτός. Δηλαδή μας είπε ότι δεν πρόκειται για τη μαφία, ε, η οποία πήγαινε να ψάξει τους ε, τραπεζίτε, αλλά το αντίστροφο. Οι τραπεζίτες πήγαιναν να ψάξουν τη μαφία. Και προκειμένου λοιπόν ε, να μπορεί να διευκολυνθεί το έργο μας, θα ζητούσα και από την Προεδρία να απευθύνει ένα συγκεκριμένο και επίσημο έτοιμα στον οργανισμό σας για το θέμα να μας διαβιβάσετε όσα είναι δυνατόν, όσα στοιχεία είναι δυνατόν, για να τα αναλύσουμε και εμείς την Επιτροπή μας. Γιατί ξέρετε ότι αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις εργασίες μας. Ευχαριστώ κύριε Μπορκέτσα. Πριν να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια ερώτηση και στους δύο. Συμφωνώ με όσα προπτάθηκαν από τον κύριο Μπορκέτσο. Πολλές φορές οι συνάδελφοι υπογράμμισαν την αναγκαιότητα από τη δική σας πλευρά να φτάνουν σε εμά ε, επιχειριακού χαρακτήρα συμβουλές. Εμείς πραγματικά καθώς ε, εδώ και λίγο καιρό υπάρχει αυτή η επιτροπή. Πραγματικά χρειαζόμαστε οι εκπρόσωποι των οργανισμών που καθημερινά δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, νομιμοποίησης παράνομων εισόδων κτλ. Να μας πείτε εσείς με ποια νομοθετικά εργαλεία, ποια νομοθετικά μέσα χρειάζεστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσετε να αυξήσετε αυτή την δραστηριότητα καταπολέμησης. Και να σας ρωτήσω κυρία Με, ε, σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία σε επιχειρησιακό, σε ερευνητικό επίπεδο έχουν γίνει πολλά. Όμως ε, είναι αλήθεια ότι κάθε έτος ε, ε πραγματικά οι κατασχέσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με το συνολικό ποσοστό της διακίνησης των ερωτικών. Έτσι λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο τι θα ήταν δυνατό να γίνει. Το ρώτησε και ο κ. Μπρουσέλινο, ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής πρόληψης και κυρίως αν ε, οι πολιτικές, όχι κατασταλτικές πολιτικές, έχουν δώσει κάποια αποτελέσματα. Και να απευθυνθώ και στον κύριο Ρόσμπεκ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στη, τον πρεσμένο Οκτώβριο ένα ψήφισμα για το οργανωμένο έγκλημα και υποστήριξε το σχέδιο της Ιντερπόλ που αφορά ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο με τη Δυτική Αφρική. Χάρη και στη δική μας υποστήριξη προχωρά το σχέδιο αυτό με μια οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να μας πείτε, μπορείτε να μας δώσετε κάποια ενημέρωση για το σχέδιο αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε από πρακτική σκοπιά. Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά αυτής εδώ της Επιτροπής πρακτικά για να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ Interpol και Europol. Θα δώσω τις εκλεπτά στον καθένα σας, καταρχήν στην κυρία Μέ και κατόπιν στον κύριο Ρόσπαχ. Παρακαλώ. Thank you again. Ευχαριστώ και πάλι. Αδιαφέρουσα ερώτηση. Έχω τον νου το χρόνο όμως. Για να απαντήσω στο συνάδελφο από τις κάτω χώρες. Είναι πολύ γενικό το θέμα του ξεπλήματος παράνομου χρήματος. Μιλάμε εδώ για τη διαφάνεια του δημοσιονομικού συστήματος. Στην πηγή πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα, να δούμε δηλαδή πώς λειτουργεί το δημοσιονομικό σύστημα να αναλύσουμε ποια είναι τα έσοδα που χρησιμοποιούν οι εγκληματικέ οργανώσεις για να μπουν στο τραπεζικό σύστημα. Και έτσι έρχομαι και στο δεύτερο σημείο που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε και ως Ευρώπη μπορείτε να κάνετε κάτι εδώ. Αλλά είναι και κάτι που αφορά το διεθνές σύστημα γιατί όλοι εσείς, οι χώρες σας, συμμετέχετε στο διεθνές σύστημα. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη γνώση. Δυστυχώς ακόμα γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα, έχουμε ελάχιστα δεδομένα, ελάχιστη πληροφόρηση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα και το τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Για να βοηθηθούμε λοιπόν, εσείς ως Επιτροπή για παράδειγμα, πρέπει να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα το ευρωπαϊκό σύστημα, ώστε να συλλέγει πληροφορίες, να αναλύει τις πληροφορίες που συλλέγει και από εκεί και πέρα ως παίχτες μέσα στο διεθνές σκηνικό να στηρίξετε και άλλες χώρες προκειμένου και αυτές να συλλέγουν δεδομένα και βέβαια να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Το θέμα της πρόληψης τώρα. Ναι, μα οι στατιστικές μας ε, το λένε κατά πόσο λειτουργεί η νομιμοποίηση ή όχι. Οπότε, ναι, έχουμε κάποια στατιστικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι ελεγχόμενες ουσίες σκοτώνουν πολύ λιγότερους από ότι οι μη ελεγχόμενες ουσίες. Το μηνόπνευμα, για παράδειγμα, ή ο καπνός. Έχουμε 5 με 7 εκατομμύρια ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας της χρήσης αυτών των ουσιών. Με τα ναρκωτικά δεν έχουμε πολύ μεγάλη βεβαιότητα, αλλά δεν είναι πάνω από 250.000. Πράγμα το οποίο δείχνει πώς επηρεάζεται η υγεία. Αυτά τα στατιστικά δεδομένα έχουμε. Αλλά μπορούμε να ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάσταση αν το σύστημα ήταν διαφορετικό. Ε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, ε, ας κάνουμε το πείραμα και μετά μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν γίνεται αυτό. Η πρόληψη, πάντως, είναι ένα πολύ καλό στοιχείο. Εμεί κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε εδώ. Δουλεύουμε σε πολλού και διάφορους τομείς. Ε, Μπορεί ανθρώπων, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία. Στηρίζουμε τα νομικά συστήματα των διαφόρων χωρών και έχουμε ένα σύστημα field offices, αξιωματούχων δηλαδή επιτόπου, σε πάρα πολλές χώρες. Διευκολύνουμε επίσης και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων που ίσως είναι λιγότερο πρόθυμες να περάσουν σε διάλογο με άλλες χώρες. Ναι, ναι, ξέρω ότι περνάει ο χρόνος. Ε, τελειώνω με τη δικιά σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Για αυτή την ε, επιχειρησιακή πρόταση. Κοιτάξτε, σε 15 λεπτά, σε 4 λεπτά δεν είναι δυνατόν να σας ε, τα παρουσιάσω αυτά αν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Οπότε τι προτείνω, αν ενδιαφέρεται η Επιτροπή σας, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, να το δούμε μαζί, ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Η οργάνωσή μας ευχαρίστως να περάσει σε αυτήν την ε, σχέση εργασίας μεταξύ μας, ώστε να καταλήξουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο και κάτι πιο συγκεκριμένο κάποια στιγμή να προτείνουμε στην ε, Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόσκλησή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα τη συζητήσουμε αύριο στους συντονιστές, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιρρήσεις. Τέσσερα λοιπόν λεπτά στον κύριο Ρόσμπαχ. Ξεκινάω με τη συνεργασία και με τις ε, συνέπειες στην Ευρώπη. Για μένα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απόλυτο ότι το σημαντικότερο είναι να αναλύσουμε τις, τις πούμε, αχίλιες πτέρνες ε, της Ευρώπης. Νομίζω ότι εξίσου σημαντικό είναι να δούμε και τι γίνεται εκτός Ευρώπης καθότι ε, οι έλεγχοι που γίνονται είναι τελείως διαφορετικοί, ε, οι αστυνομικές αρχές, ε, αν θέλετε, αυτές που βρίσκονται στην Αφρική, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση τοποθετείται και η δική σας η ερώτηση, που έχει σχέση με την προαγωγή προγραμμάτων, περιφερειακών προγραμμάτων, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την κατάθεση εκθέσεων. Εμείς προτείνουμε και μία μεταρρύθμιση στην Europol. Προτείναμε μεταρρύθμιση και τοποθετηθήκαμε στο τι ακριβώς είναι σημαντικό κατά την άποψή μας. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, η πρόληψη είναι σημαντική και σημαίνει ότι πρέπει να διερευνηθεί πλήρως το φαινόμενο με μη κυβερνητικού οργανισμούς ε, και με άλλους ε, έτσι ώστε ε, για να εντοπιστούν οι καλύτερες, οι βέλτιστες προσεγγίσεις. Αυτή τη στιγμή μας στηρίζουν ουσιαστικά οι Καναδοί στην Αμερική στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουμε στην Αμερική. Άρα δηλαδή να υπάρχει συνδυασμός εκπαίδευσης επιτόπου με τις άμεσα ενδιαφερόμενες αρχές, να βρισκόμαστε όλοι ε, και αφού γίνεται εκπαίδευση να έχουμε ως στόχο και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μετά δηλαδή την εκπαίδευση να γίνεται και επιτόπου μια επιχείρηση όπου θα αποδεικνύεται το τι μάθαμε, αν δηλαδή ήταν αποτελεσματική η άσκηση. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό για να εντοπίσουμε καλύτερα την αλλαγή των διαδρομών, την αλλαγή των ε, μέσων που ε, χρησιμοποιούν ε, οι συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος και βέβαια με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και άλλων. Όσον αφορά τώρα τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, τα ηλεκτρονικά μάλλον εγκλήματα. Η Europol, η ε, Interpol συνεργάζονται στενά. Η Europol θα οργανώσει το Ευρωπαϊκό Όργανο του Κυβερνοχώρου και εμείς έχουμε μια ειδική μονάδα στη Σιγκαπούρη που θα βοηθήσει, ε, γιατί οι πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Τώρα, όσον αφορά στην ε, συνεργασία την οποία προάγει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω το πρόγραμμα ΒΑΠΙΣ σε σχέση με τη Δυτική Αφρική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και ακούσαμε το ρόλο που παίζει αυτή η περιοχή σε αυτό το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σημαντικά μέτρα ε, που εφαρμόζουμε, μέτρα πρόληψης, αλλά να είναι και διάρκειας Έχουμε και συγκεκριμένες αποστολές σε, τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες επιτόπου διαπιστώνουν ε, κατά πόσον διατηρείται η αναμενόμενη ποιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, ε, για την σαφήνεια με την οποία μιλήσατε και για την προσφορά συνεργασίας. Ε, αυτό είναι κάτι που θα το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας και θα ξανασυνεργαστούμε για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτές τις προτάσεις λοιπόν ε, θέλω να σας αποχαιρετήσω και πάλι ευχαριστώντας σας για τη δουλειά σας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχε προβληθεί ε, να ε, κλέξουμε τον τέταρτο αντιπρόεδρο γιατί παρετήθηκε ο προηγούμενος Mm. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις, να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ε, βουλευτές ε, σε αυτή την επιτροπή για να μπορείτε να εκλέξετε έναν αντιπρόεδρο. Κύριε Σόντεργαρτ δεν ξέρω αν έχετε Κύριε Σόντεγκαρτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να προτείνω τον Ντένις Τιγιόν από την δική μας την ομάδα ως αντιπρόεδρο και ελπίζω να γίνει αποδεκτή η υποψηφιότητά του. Ο υποψήφιος δέχεται την υποψηφιότητα. Άλλοι επιθυμεί κάποιος άλλος να θέσει υποψηφιότητα. Ματιέ, θέλετε να παρέμβετε, να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά πρόκειται για πολιτική συμφωνία, δεν θα φέρουμε αντίρρηση λοιπόν. Ήθελα να πω όντως ότι ο κύριος Ντεγιόνκ αρχίζει άσχημα τη θητεία που του ε, προσέφερε η διάσκεψη των Πρόεδρων γιατί αναφέρθηκε ε, στην ομοποίηση της κάναβης και για μας ε, δεν είναι καθόλου αποδεκτό κάτι τέτοιο, κυρίως σε μια επιτροπή όπως η δική μας. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Πρέπει εγώ να ρωτήσω τον υποψήφιο που έχει διδεκτεί την υποψηφιότητα αν έχει συμπληρώσει τη δήλωση σχετικά με ε, τα οικονομικά συμφέροντα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μου λέει η γραμματεία ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Δεν ε, έχει ζητηθεί λοιπόν ψηφοφορία μυστική. Έτσι λοιπόν ε, εκλέγεται ο υποψήφιος. Καλό λοιπόν ε, τον ε, Αντιπρόεδρο Ντεγιόν και να καθίσει εδώ δίπλα μου. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο πάνελ, στη δεύτερη ομάδα. Ο τίτλος ε, εδώ είναι παράνομη διακίνηση και παραποίηση. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα μια παρουσίαση μιας κοινή τηλεοπτικής επιχείρησης, μιας επιχείρησης που οργανώθηκε από την ΟΛΑΦ με την υποστήριξη της Europol σχετικά με τα παραποιημένα αγαθά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρέμβαση για να εμβαθύνουμε και σε μια σειρά πτυχών που ήδη είδαμε στην Επιτροπή μας, δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών αρχών. Και έχουμε εδώ τον κύριο Χιτερή από την Όλαφ και τον Κρίς Βαστιχίτς από τη Γεροπόλ θα έχουμε μια κοινή παρουσίαση και θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων ε, με ε, τον εκπρόσωπο της Γραμματείας του Συμβουλίου, τον κύριο Τζένσον, ε, σε σχέση με την εμπειρία της Μόνιμης Επιτροπής για την Ασφάλεια, την ΚΟΖΗ, για τη συνεργασία στον τομέα της διακίνησης και της περαποίησης. Και πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΚΟΖΗ, θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικός ρόλος αυτός και θα πρότεινα να οργανωθεί συζήτηση ως εξής. Καταρχήν, να ακούσουμε στους εκπροσώπους της Όλαφ και της Europol. Έχετε στη διάθεσή σας και οι δύο, δέκα 12 λεπτά το πολύ και κατόπιν ο κύριος Γκένσον θα έχει στη διάθεσή του 15 λεπτά. Έτσι λοιπόν ε, θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος ερώτα-απαντήσεων με προτεραιότητα ο εισηγητής και οι συντονιστές, δύο λεπτά, κατόπιν θα απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας και αν υπάρχει χρόνος θα έχουμε ένα νέο γύρο ερώτα-απαντήσεων. Να δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στον κύριο Τεριχέν για την ΟΛΑΦ 10-12 λεπτά το πολύ παρακαλώ έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η ΟΛΑΦ έχει ως πεδίο δράσης για την πνευματική διοκτησία περιορίζεται στην εισαγωγή, την εξαγωγή και το τράνζιτ με τρίτε χώρες. Στόχος δηλαδή δεν είναι να καλύψουμε εδώ την εσωτερική αγορά. Η δράση μας εγγράφεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπάρχουν μέτρα τα οποία υιοθετούνται από την TaxUD, από τη Γενική Διεύθυνση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον έλεγχο και την ε, παρέμβαση, αλλά υπάρχει και ένα πλαίσιο καταπολέμηση τη απάτης που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση τάξη. Πρόκειται για τον κανονισμό 1383 του 2003. Στο άρθρο 22 συγκεκριμένα μιλάει για την καταπολέμηση της απάτης. Η διάταξη αυτή λοιπόν μας επιτρέπει να κάνουμε διοικητικές ανακρίσεις αλλά και να επιβλέπουμε τι κάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά τη διακίνηση την αποθήκευση υλικού. Υπάρχει συμφωνία επίσης αμοιβαία αρρωγή με τρίτες χώρες και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιε διοικητικέ έρευνες με τη συνεργασία των τρίτων αυτών χωρών στις τρίτες χώρες. Κάτι το οποίο συμπληρώνει βέβαια τη δράση ε, των συναδέλφων από την Europol και την Eurojust. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα δράσης όπου καταφέραμε να έχουμε συνεργασία όχι μόνο με τις αρχές τρίτων χωρών, αλλά και γενικότερα με τρίτες χώρες, αλλά και με την Ευρωπόλ και την ε, Ιντερπόλ. οι δράσεις αυτές συντονίστηκαν από εμάς και πρόκειται για την δράση Σιρόκο στην Νότια Ευρώπη. Έχουμε ένα επιχειρησιακό κέντρο λοιπόν, το οποίο χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες δράσεις που περιορίζονται σε δύο ή τρει εβδομάδες το πολύ. Βασιζόμαστε σε ένα σύστημα πληροφορικής ιδιαίτερα ισχυρό, το οποίο συνδέει διάφορους φορείς σε τρίτες χώρες αλλά και στις χώρες μέλη και όπου έχει πρόσβαση και η Interpol και η Europol όσο καιρό διαρκεί. Ο συντονισμός γίνεται από την Όλαφ με μία εφαρμογή πληροφορικής, την μονάδα εικονικού επιχειρησιακού συντονισμού. Βλέπετε εδώ ότι συμμετέχουν 27 χώρες όπως και τα τελωνία και οι συνάδελφοι από την ε, ταξίτ. Χρησιμοποιούμε 13 αξιωματούχους επιτόπου και συμμετέχουν και η Αιγύπτος, το Μαρόκο και η Τουρκία. Πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μαζί τους ήταν εξαίρετη. Βάσει λοιπόν ενός επιχειρηματικού σχεδίου που καθορίζει ο ΛΑΦΕΚ των προτέρων με κριτήρια Ζητήθηκε για διάφορα παραποτοκιβώτιο από 11 χώρες της Μεσογείου αλλά και τις 27 χώρες μέλη, ζητήθηκε να συλλέξουν στοιχεία και συνέληξαν στοιχεία για μια περίοδο 10 ημερών στοιχεία για διάφορα ύποπτα εμπαρευματοκιβώτια. 411. Εδώ βλέπετε από την Κίνα ή από τα Αραβικά ε, Εμμυράτα που για μας είναι ευαίσθητες περιοχές και είδαμε τι έγινε και με τη μεταφόρτωση από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη μέσω είτε τα Ραβικά Εμμυράτα είτε μέσω κάποιας χώρας της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Στόχος μας ήταν να δούμε τι γίνεται με πλαστά ε, σιγαρέτα ή με λαθρεμπόριο γνήσιων σιγαρέτων. Τα λιμάνια επιλέχθηκαν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που καθορίστηκαν εκ των προτέρων. Η δράση αυτή αποτελείται από διάφορα στάδια το επιχειρησιακό στάδιο ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου του 2010 και ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου του 2010. 411 μετακινήσεις ύποπτες εντοπίστηκαν από, τα, από τις επαφές μας. Τελικά επιλέξαμε 300 ύποπτα παραβατοκιβώτια όταν στενέψαμε κάπως τα κριτήριά μας. Η Europol λοιπόν και η Interpol είχαν ε, άμεση πρόσφαση στις πληροφορίες και διασταύρωσαν με τις δικές τους αναλύσεις και είδαν από τα 411 παραπτωκιβώδια 77 Όντω η Γεροπόλο τα είχε ψάξει ακόμα και αν δεν είχε καταλήξει όσον αφορά τις δραστηριότητε σχετικά με πλαστά αγαθά, αλλά μπορεί να πρόκειται και για νομοποίηση παράνομου χρήματο είτε για ε, παρανομοχήματα. Το αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν ε, ότι κατασχέθηκαν 40 από τα 300 τα οποία ψάξαμε. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα 35 εκατομμύρια σιγαρέτα για παράδειγμα κατασχέθηκαν. Όπως ε, επίσης είχαμε και δύο περβατοκιβώτια με καπνό για στριχτά τσιγάρα. 1071 ε, κιλά. Αλλά βρέθηκαν και άλλες ε, τσάντες με πλαστά προϊόντα, είτε πρόκειται για ρούχα, είτε για παπούτσια, τσάντες, παιχνίδια, ηλεκτρονικό υλικό αλλά επίσης και κατασχέθηκαν, κατασχέθηκε ένα βαρματοκιβώτιο με 7.038 λίτρα ε, αλκοολούχων ποτών μη δηλωμένων και συλλήφθησαν τρία άτομα. 8 εκατομμύρια ευρώ είναι η απώλεια από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Ετοιμάστηκε καλά λοιπόν η δραστηριότητα αυτή και συνεργαστήκαμε και με τους συναδέρφους από την Μάλτα για μια άλλη ε, διοικητική έρευνα όπου κατασχέθηκαν 8 εμπορματοκιβώτια από τα Ενωμένα Εμμυράτα προς την ε, Μάλτα. Και είχαν μέσα είτε ψυγεία είτε στότερ, τόστερ και διαπιστώσαμε, έτσι μάλλον δήλωναν, και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για φάρμακα μέσα σε καταψύχτες βρήκαμε διάφορα φάρμακα. Επρόκειτο και εδώ για τσάντες, πίκνικ που είχαν μέσα τέτοια προϊόντα. Και μέσα στις τοστιέρες επίσης βρήκαμε τραμαντόλ, που είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται για να ανακουφίζει από τον πόνο και το χρησιμοποιεί ο ιατρικός κόσμος. 118 εκατομμύρια καψούλες βρήκαμε στα 8 εμπαρματοκιβώτια τα περισσότερα με πρεμαντόλ. Η άδεια έτσι και αλλιώς έχει εκπνεύσει, πράγμα που σημαίνει ότι κυκλοφορεί ελεύθερα το προϊόν αυτό. Επειδή όμως υπήρχε λανθασμένη δήλωση και ήταν κρυμμένα τα προϊόντα αυτά, κατασχέθηκαν τα προϊόντα αυτά με άλλης νομικής βάσης. 8 εκατομμύρια πάντως ε, ταμπλέτες άλλου φάρμακου κατασχέθηκαν επειδή ήταν πλαστά. Είναι σημαντικό εδώ να γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε και κανένα επεξηγηματικό σημείωμα οδικής χρήσεως δηλαδή για τα προϊόντα αυτά. Οι ποσότητες εξάλλου δεν ανταποκρίνονται βέβαια και στις ανάγκες των ε, ε, νοσοκομείων στη Λιβύη όπου προορίζονται. Οπότε από τις επαφές που είχαμε και με την Αίγυπτο, όπου και εκεί επρόκειτο να καταλήξουν τα φάρμακα, ε, καταλάβαμε ότι έπρεπε να κατασχεθούν και βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εμποδίζει τις κατασχέσεις σε περίπτωση τράνσιτ είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ε, συζητάμε για τις πληροφορίες αυτές με τις διαφερόμενες τρίτες χώρες για να έχουμε από αυτές όλες τις σχετικές πληροφορίες. Πώς ε, προχωράμε τώρα. Η γενική μας διεύθυνση θέλει επιμονή μου βάσεως να έχουμε τέτοιες δράσεις με αξιωματούχου σύνδεσης οι οποίοι είναι κατεστημένοι στις χώρες μέλη και σε συνεργασία και με κάποιον από την Europol. Επίσης προβλέπουμε να τροποποιήσουμε τον ε, κανονισμό που διέπει τις δραστηριότητές μας έτσι ώστε και η Europol να μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές προς το παρόν. Έχει πρόσβαση μόνο σε μία βάση ε, δεδομένων για τις ε, κοινέ αρμοδιότητες και όχι τις επιμερισμένες δηλαδή και όχι και τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Europol, στον Κρίς Βάλστακιστ, για να σύγχυσε να μας μιλάει για αυτή την κοινή τελωνιακή επιχείρηση μεταξύ ΟΛΑΦ και Europol. Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί ακροτέ, είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα να βρίσκομαι εδώ εκ μέρου της Europol για να σα ενημερώσω όσον αφορά το φαινόμενο αυτό της ε, πειρατεία προϊόντων, των πλαστών ε, προϊόντων και της παραχάραξης και τι κάνουμε στην Europol για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Μιλάμε λοιπόν για τα πλαστά προϊόντα, τα πειρατικά. Ο καθένας έχει στο μυαλό του διάφορα είδη πολυτελεία. αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτά. Στην πραγματικότητα ζηλεύω μερικές φορές του συναδέρφους από τη μονάδα καταπολέμησης λαθρεμπορίων ναρκωτικών ή άλλους, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν και έχουν σύντομα αποτελέσματα. Όταν πρόκειται για πλαστά όμως προϊόντα είναι πολύ πιο δύσκολο να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στις δικές μας δραστηριότητες. Είτε πρόκειται για την αστυνομία, είτε πρόκειται για τη δικαιοσύνη, γιατί βλέπετε τι λένε, ε, για λίγα πλαστά ρούχα τώρα εμείς δεν θα ξεκινήσουμε μια ολόκληρη δράση. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλο πρόβλημα. Άρα βλέπετε ότι το εμπόδιο είναι η νοτροπία πολλές φορές. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για προϊόντα πολυτελείας. Η τελευταία τάση τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται είναι ότι αλλάζει το τοπίο. Περνάμε σε προϊόντα καθημερινής χρήσης είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε πρόκειται για ξηρά φάκια ή ξηριστικέ μηχανές, είτε για στυλό, είτε για απορριπαντικά, μπαταρίες κλπ. κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και έχει να κάνει με την υγεία, την ασφάλεια και τελικά πώς δρούν ε, εγκληματικές οργανώσεις και πώς εμπλέκονται στο εμπόριό μας. Αυτό είναι και ο λόγο για του οποίου η Europol δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα προσπαθώντα να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Το 2008 φτιάξαμε μια ομάδα, μια μονάδα δηλαδή, η οποία έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό των πλαστών προϊόντων και της πειρατείας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν νέε τάσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή περνάμε από τα προϊόντα πολυτελείας στα προϊόντα καθημερινή χρήση. Υπάρχει επίσης και μια άλλη αλλαγή, αν κοιτάξουμε τι γίνεται με τα φάρμακα. γιατί περνάμε από το lifestyle drugs στα life saving drugs, δηλαδή από τα απλά προϊόντα ε, φαρμακευτικής χρήσης περνάμε σε φάρμακα τα οποία είναι πολύ αναγκαία για να σώσουν τη ζωή ορισμένων ανθρώπων, είτε πρόκειται για το, τη λευχαιμία, είτε άλλα. Μέχρι τώρα ξέραμε για τα διάγκρα ή για άλλα, αλλά τώρα περνάμε, όπως σας είπα, και για φάρμακα τα οποία κανονικά σώζουν ζωές. Ερευνούμε λοιπόν το θέμα και διαπιστώνουμε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις τελικά έχουν παρελθόν από λαθρεμπόριο άλλων προϊόντων. Πρόκειται δηλαδή για μία business η οποία αποφέρει πολλά σε αυτούς, κακά τα ψέματα. Δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά κλιματικέ οργανώσει επειδή τη βρίσκουν ωραία και ευχάριστη, αλλά γιατί καταλαβαίνουν ότι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά από αυτήν. Ξέρω ότι μου έχετε δώσει λίγο χρόνο και έχω κακή φήμη, συνήθω δεν τηρώ το χρόνο μου, προσπαθώ όμω. Γι' αυτό και θα επικεντρωθώ σε δύο φαινόμενα με τα οποία ασχολείται η Europol. Το ένα είναι τα παρασιτοκτόνα και το άλλο είναι τα πλαστά φάρμακα. Για τα παρασιτοκτόνα πρώτα. Είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Αν δείτε λοιπόν τις στατιστικές του 2009, 100 τόνους είχαμε κατασχέσει. Το 2011 3.000 τόνοι. Έτσι λοιπόν, ασχολήθηκα κι εγώ λιγάκι με τα παρασιτοκτόνα και την κατάσχεσή τους. Τι σημαίνει ένας τόνος. Πρόκειται για υγρά, έτσι. Με ένα τόνο μπορείτε ε, ολόκληρο το δουκάτο του Λουξεμβούργου να καλύψετε. Για να καταλάβετε δηλαδή για τι ποσότητες μιλάμε είναι συνεπώς ε, νούμερα το οποίο μιλάνε από μόνο τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 3.000 τόν τι σημαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ότι με τα πλαστά παρασιτοκτόνα μέσα βάζουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και καταλαβαίνετε ότι να βλέπετε εδώ πέρα στα slides τις ε, διαφάνειες, τις καλλιέργειες, οι οποίες βέβαια καταστρέφονται τελικά. Και ίσως αυτό να είναι το πιο απλό, γιατί αυτά τα φυτά που βλέπετε εδώ δεν ε, δίνουν καρπούς που θα φάμε αργότερα. Υπάρχει όμως και άλλο πρόβλημα με τα παρασιτοκτόνα είχαμε την Flashpoint που ήταν μια επιχείρηση. Να, εδώ πέρα από το Πεκίνο έρχεται μια, ένα επιβατικό αεροπλάνο. Περνάει από τη Βουδαπόστη. Από τη Βουδαπέστη λένε, ο, ακούμε, έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχουν ε, ναρκωτικά. Ψάχνουμε το αεροπλάνο, δεν τα βρίσκουμε. Βρίσκουμε όμως τέσσερις τόνους παράνομα παρασιτοκτόνα. Μετά την ε, ανάλυση διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για χημικές ουσίες που έμειναν σε μια θερμοκρασία 24 βαθμών. Αυτό Δεδομένου ότι οι ουσίες αυτές είναι επικίνδυνες, καταλαβαίνετε ότι έχουν και μια άλλη επικινδυνότητα για τους επιβάτες δηλαδή του αεροπλάνου, γιατί σε αυτήν την θερμοκρασία οι ουσίες αυτές γίνονται πολύ πιο επικίνδυνες. Τώρα για το φάρμακο έγκλημα. Με την Γενική Διεύθυνση Τάξου του συνεργαζόμαστε εμείς και είδαμε το 2008 6,5% των υποθέσεων που είχαν να κάνουν με τα πλαστά φάρμακα και 5% ήταν οι κατασχέσεις για 9 εκατομμύρια. Το 2009 είχαμε φτάσει στο 8% έρευνες και 10% κατασχέθηκαν ε, προϊόντα αξίας 11 εκατομμυρίων. Το 2010 έγινε πάλι κατάσχεση 25 εκατομμυρίων ευρώ αξίας ε, φαρμάκων. Τα τρία ήταν είτε για ορολιμόξεις, είτε αντιφλεγματόδη, είτε για καρδιακές παθήσεις. Το 2011 532 διαφορετικά είδη πλαστών φαρμακευτικών προϊόντων κατασχέθηκαν. Και το 2008 είχαμε πλαστά φάρμακα που εντοπίστηκαν σε 118 χώρες. Το 2009, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ανισχυτικό, είναι ότι είχαμε 536 περιπτώσεις όπου διαπιστώσαμε ότι πλαστά φάρμακα είχαν μπει στο νόμιμο δίκτυο κυκλοφορίας φαρμάκων, στη χοντρική δηλαδή. Εδώ βλέπετε ποια είναι η τάση όσον αφορά το φαρμακό έγκλημα. Τι έχει γίνει δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια. Και εδώ βλέπουμε ότι τα περισσότερα τα έχουμε στην Ασία. Αλλά αν κοιτάξετε και την Ευρώπη, διαπιστώνετε ότι έχουμε 351 περιπτώσεις. Συνολικά είναι κάπου 2.000 οι περιπτώσεις σε όλες τις υπήρους. Εδώ βλέπετε όλες τις υπήρους που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις πλαστών ε, φαρμάκων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτές ε, παράγουν κάποια πλαστά για τον καρκίνο, για παράδειγμα. Τώρα όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας. Μια από τις πιο πρόσφατες όπου συμμετείχε η Europol ήταν η Τρίμπουλης. Έχει γίνει η σχετική ανάλυση και συντονισμός μεταξύ μας. Στη Χάγη γίνεται ο συντονισμός. Η Γουάρδια Σεβίλα από την Ισπανία συμμετείχε και η MHRA από το Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν αντίστοιχε επιχειρήσεις και τελικά συνελήφθησαν έξι άτομα, τέσσερα στην Ισπανία, δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνολικά είχαμε 300.000 δόσεις πλαστών φαρμάκων που κατασχέθηκαν. Και πάγωσαν βέβαια και τα περιουσιακά στοιχεία σε διάφορους τραπεζικούς οργανισμούς, κατασχέθηκαν και κινητά και υπολογιστές. Άλλες δράσεις είναι η όψων, για παράδειγμα, σε συνεργασία ανάμεσα στην Europol και την Interpol. Είναι μια μεικτή λοιπόν επιχείρηση μεταξύ μας. Μέσα σε μια εβδομάδα δηλαδή επικεντρωθήκαμε σε πλαστά τρόφιμα και ποτά. Πάνω από 700 τόνοι τροφίμων και ποτών κατεσχιάθηκαν σε 11 διαφορετικές χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Τέλος, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Συνεργαζόμαστε εντατικά. Interpol, Eurojust, ε, Olaf και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία αυτή. Υπάρχουν επιχειρήσεις τις οποίες ήδη συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι το έγκλημα δεν σταματάει στα σύνορα, άρα γι' αυτό η Europol, η Interpol και άλλες οργανώσεις όπως η Olaf πρέπει να συνεχίζουν και να μην σταματάνε στα σύνορα. Μια άλλη επιχείρηση τώρα στην οποία δραστηριοποιούμεθα με τα παρασιτοκτόνα έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Και γιατί, γιατί είναι ένα περίπλοκο θέμα. Ε, υπάρχουν πολύ άγνωστοι παράγοντες. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε πρώτα περισσότερα, να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, να ενημερωθεί η αστυνομία και άλλες οργανώσεις πριν προχωρήσουμε σε επιχείρηση. Φέτος λοιπόν έχουμε οργανώσει ένα σεμινάριο με την Eurojust, την Europol, την Olaf, ώστε να βαθύνουμε περισσότερο στο θέμα των παρασιτοκτόνων. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε επιτυχή αποτελέσματα της αστυνομίας μας και των τελωνίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh, e Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, εμπεριστατωμένη ανάλυση και θα ήθελα να δώσω το λόγο για 15 λεπτά στον ε, εκπρόσωπο της Γραμματείας του Συμβουλίου, τον κύριο Γκένσον, ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για τις εμπειρίες που έχει κάνει από τις ε, επιχειρήσεις που αναπτύσσει η Κόζη, ε, κυρίως με ειδική αναφορά στη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το ρόλο που παίζει η Κόζη στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών και της παραποίησης. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Πώς, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για την κόζη. Εγώ δεν έρχομαι από ε, την ε, επιχειρηματική μονάδα. Έχω περισσότερο επιχειρησιακή εμπειρία και προσπαθούμε να χαράξουμε πολιτική και να διευκολύνουμε ε, τα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας. Η ΚΟΖΗ, η Επιτροπή Ιστορικής Ασφάλειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια νεόκοπη Επιτροπή προέκυψε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και προέκυψε μετά από συζητήσεις που έγιναν στην ομάδα εργασίας 10, η οποία τότε ε, είχε ως ε, επικεφαλής τον κύριο Μπρούτον και κατέστησε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαζόταν ένα είδος ειδική μονάδα, ειδικού φορέα, για να εργάζεται σε θέματα συντονισμού στην εσωτερική ασφάλεια. Τότε λοιπόν είχαμε ε, δύο μονάδες στην Σκύφα για ε, το άσυλο και το άρθρο 36 που ασχολείται με την συνεργασία των αστυνομικών αρχών και των ε, αρχών δικαιοσύνης. Καμία όμως από τις δύο δεν ασχολείται με, την, ε, με τον καθημερινό συντονισμό. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο Τάμπερε οδήγησαν στη σύσταση μιας Επιτροπής αρμόδιες για τις αστυνομικέ αρχές κατέστησε σαφές αυτή η ομάδα δράσης δεν ήταν το κατάλληλο όργανο για να αντιμετωπίσει θέματα συντονισμού. Ποια ήταν λοιπόν η λύση να συσταθεί ένας νέος οργανισμός ε, που βασίζεται στο άρθρο 71 της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι το φόρουμ εκείνο που ασχολείται με θέματα συντονισμού εσωτερικής ασφάλειας. Η Επιτροπή ήταν σαφώς απόφαση του Συμβουλίου. Μία νεοκόπη λοιπόν Επιτροπή. Ε, τώρα ποιος συμμετέχει. Προφανώς όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Κροατίας ως παρατηρητής. Επίσης έχουμε και τις χώρες που συμμετέχουν στην μεικτή επιτροπή με τις συμφωνίες Σέγκεν. Δηλαδή, κάθε φορά ε, που ασχολούμεθα με θέματα του Σέγκεν, Νορβηγία, Ισλανδία, ε, Ελβετία και Λίχτενστάιν ε, συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Έχουμε την επιτροπή και όλους τους φορείς που ασχολούνται με θέματα εσωτερικής ασφάλειας Europol, Eurojust, ιδιαίτερα αυτήν, γιατί η εσωτερική ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα των αστυνομικών αρχών, αλλά και της συνεργασίας για θέματα ποινική δικαιοσύνης. Συμμετέχει λοιπόν η Eurojust, η Frontex για θέματα εξωτερικών συνόρων, η CIPOL για την εκπαίδευση, η CCDMA, μια ειδική μονάδα που ασχολείται με τα ναρκωτικά, Όλαφ και επίσης η Interpol εφόσον έχουμε θέματα τα οποία την αφορούν δηλαδή που έχουν σχέση με τις ε, εξωτερικές σχέσεις και σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν τη συμμετοχή όλων αυτών των φορέων της εσωτερικής ασφάλειας είτε ε, σε επίπεδο κρατών μελών είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορείς λοιπόν ε, συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες και έχουν τη δυνατότητα μέσα από το φόρουμ να συντονίζουν όλα τα προγράμματα που οργανώνει η Επιτροπή. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Τώρα, για τα συγκεκριμένα θέματα, την εμπειρία της Κόζια και τη συνεργασία ε, στον τομέα της διακίνησης και της παραποίησης. Λίγα μόνο είναι τα προγράμματα που ασχολούνται με θέματα αυτά. Όμως υπάρχουν αρκετά προγράμματα όπου έχουμε άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις με την διακίνηση και την παραποίηση. Θα σας παρουσιάσω όλα αυτά τα προγράμματα που ελέγχουμε εμείς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που εισήχθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009 και αυτό καλούσε το να υπάρξει μια μονάδα ιστορικής ασφάλειας. Και μια προτεραιότητα της ΚΟΖΗ είναι να ελέγχει ε, την ε, στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Η στρατηγική αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεσπίστηκε το 10 υπό την σχετική προεδρία δανική και το οργανωμένο έγκλημα αντιμετωπίστηκε ως μια βασική αλλαγή ε, σε σχέση με την ιστορική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή λοιπόν τη στρατηγική η διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων, ε, όπλων, η παραποίηση αυτά προφανώς έχουν άμεση σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, αυτά αντικατοπτρίζονται και στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας της ε, ΚΟΖΗ, το οποίο συστάθηκε υπό την Βελγική Προεδρία το 2010, με στόχο η ΚΟΖΗ ε, να ε, έχει ένα πρόγραμμα για, τις, τρόικα, για την Τρόικα που θα ακολουθούσε. Ορίστηκε λοιπόν το πρώτο πρόγραμμα στο πλαίσιο της δουλειάς της Τρόικα. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα θέματα, το πρώτο που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οργανωμένο και το σοβαρό έγκλημα. Το δεύτερο έχει σχέση με ναρκωτικά. Έχουμε δύο συμφωνίες για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Πρώτο η ηρωίνη κοκαίνη, δεύτερον για συνθετικά ναρκωτικά. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσω με την ευρωπαϊκή πολιτική για το οργανωμένο και το σοβαρό έγκλημα. Αυτή η πολιτική ανάγεται σε μια Βελγική στρατηγική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 9-10 και εγκρίθηκε τέλος του 2010 Βελγική ήταν η πρωτοβουλία και το πρόγραμμα έφερε τον τίτλο «Αρμονία». Η ιδέα λοιπόν ήταν να ε, οριστούν οι προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτή λοιπόν η πολιτική ορίστηκε το 2010 και σήμερα αποτελεί τη βάση της δουλειάς της ΚΟΖΗ στον τομέα του οργανωμένου και του σοβαρού εγκλήματος. Η πολιτική αυτή προσπαθεί να διαμορφώσει έναν πολιετή κύκλο και μία σαφή μέθοδο για να εφαρμόζονται και να αξιολογούνται οι προτεραιότητες στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Πάντα έχοντας κατά νου το οργανωμένο έγκλημα και το σοβαρό διεθνές έγκλημα. Συμφωνήσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ε, με συγκεκριμένες πολιτικές για την περίοδο 11 έως 13 με βάση την ε, αξιολόγηση απειλών του 2011 όπως την ε, παρουσιάστηκε Europol. Μετά από αυτές τις δύο περιόδους θα έχουμε μια τετραετή πολιτική από το 13 μέχρι το 17 που θα βασίζεται στην αξιολόγηση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα επανέλθω αργότερα για το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα για την αξιολόγηση των απειλών. Η μεθοδολογία λοιπόν επιτρέπει στο ε, Συμβούλιο να συμφωνήσει σε κοινέ ε, προτεραιότητες ε, έτσι ώστε να εστιάσει καλύτερα την προσοχή του στο οργανωμένο έγκλημα. Με βάση λοιπόν την αξιολόγηση των απειλών. Από το Europol του 2011, το Συμβούλιο συμφώνησε σε οκτώ προτεραιότητες στον αγώνα κατά του οργανωμένου κλίματο για την περίοδο 2011 μέχρι 2013. Πρώτη προτεραιότητα αφορά την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων ομάδων που βρίσκονται στη Δυτική Αφρική και σχετίζονται με κοκαίνη και ηρωίνη που τη μεταφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη προτεραιότητα έχει σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια έτσι ώστε να αμβληνθεί ο ρόλος αυτής της περιοχής ως ε, βασικό κλειδί για την διακίνηση ναρκωτικών. Ε, είναι ένα κέντρο σοβαρό, ε, κυρίως με επίκεντρο την Αλβανία η τρίτη προτεραιότητα που ορίστηκε σε αυτόν τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων των οργανωμένων εμάδων που διευκολύνουν την παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως με ε, λαθρομετανάστες που έρχονται από την Τουρκία και από τη Μεσόγειο και από περιοχές κοντά στη Βόρεια Αφρική. Η τέταρτη προτεραιότητα, την οποία αποφάσισε το Συμβούλιο, έχει σχέση με τη μείωση της παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών ε, και νέων ε, ψυχοδιαγερτικών. Η πέμπτη προτεραιότητα έχει σχέση με την ανακοπή ε, μεταφοράς κοκαίνης, ηρωίνης, κανάβεως, παραποιημένων προϊόντων η, έξι, η έκτη προτεραιότητα αφορά την αντιμετώπιση όλων των μορφών ε, παράνομης διακίνησης ανθρώπων ε, με στόχο ειδικέ εγκληματικέ ομάδες που αναπτύσσουν τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες κυρίως στα νότια σύνορα και τα νοτιοανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβδομη προτεραιότητα έχει σχέση με την μείωση της δυνατότητας ταυτότητας ε, οργανωμένων, περιφερόμενων οργανωμένων ομάδων και τελευταία προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί ο αγώνας ε, κατά της, ε, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Αυτές λοιπόν είναι οι οκτώ προτεραιότητες που όρισε το Συμβούλιο έτσι ώστε ε, να υπάρχει καλύτερος ε, συντονισμός σε σχέση πάντα με την εσωτερική ασφάλεια. Το Συμβούλιο λοιπόν καθόρισε τις προτεραιότητές του και θέλουμε να δούμε τι συνέβη κατόπιν. Εμείς ε, θέλουμε να ορίσουμε τους βασικούς παράγοντες για κάθε προτεραιότητα. Για κάθε προτεραιότητα να υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο από το 2011 μέχρι το 2013. Μισό λεπτό. Σας διακόπτω ένα λεπτό. Έχω πρόβλημα στο πόδι και πρέπει να περπατήσω για λίγο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω ε, την ε, κυρία Ματιώ, επειδή δεν υπάρχει εδώ αντιπρόεδρος, να έρθει στο Προεδρείο να με αντικαταστήσει για λίγο. Η κυρία Ματιώ είναι μέλος της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας που συμμετέχει εδώ σε εργασίες. Για κάθε λοιπόν στρατηγικό στόχο υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης ε, το οποίο ε, πρέπει να εφαρμοστεί. Γι' αυτό το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ε, η Europol, η Frontex, η Cipol, όλες, όλοι αυτοί οι οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αν δούμε τώρα λιγάκι αυτό το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, υπάρχουν πέντε τα οποία εξετάζουν άμεσα ή έμεσα την παράνομη διακίνηση και την παραποίηση. Το πρώτο που έχει σημασία είναι το πρόγραμμα δράσης στη Δυτική Αφρική αυτό εστιάζει την προσοχή του κυρίως ε, ε, στην σαρκωτικά που έρχονται από τη Δυτική Αφρική. Το δεύτερο πρόγραμμα δράσης αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια υπό την καθοδήγηση της Ιταλίας. Εδώ βασιζόμαστε σε αυτή τη μορφή εγκλήματος. Το τρίτο πρόγραμμα δράσης έχει σχέση με την παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων υπό την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά πάμε στα συνθετικά ναρκωτικά υπό την Πολωνία και τέλος ε, ε, στην ε, εισαγωγή μέσω εμπορευματοκιβωτίων. Βλέπετε λοιπόν ότι για κάθε ένα από τα προγράμματα δράσης υπάρχει ένα κράτος μέλος ε, το οποίο αναλαμβάνει να διαχειρίζεται το πρόγραμμα, να το εφαρμόζει και αργότερα να το αξιολογεί σε συνεργασία με μας. Πρόσφατα η υπηρεσία μας ε, ε, διεξήγαγε τον συντονισμό των προγραμμάτων δράσης. Σήμερα λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει μια κάπως μεικτή εικόνα. Υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές, ε, που εντοπίζονται, ε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση, κυρίως σε σχέση με τη συμμετοχή των κρατών μελών σε τέτοιου είδους ε, προγράμματα. Ε, βεβαίως, σε σημασία και ρόλο παίζει και η χρηματοδότηση όλων αυτών των δράσεων. Ας δούμε λιγάκι ποιο θα είναι το μέλλον Έχουμε, όπως σας είπα, ένα κύκλο ε, πολιτικών από το 13 μέχρι το 17 και η βάση αυτού του κύκλου δεν είναι το ε, κλασικό οργανωμένο έγκλημα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αλλά ε, θα υπάρξει μια νέα έκθεση που θα εστιάζεται στην απειλή από το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα. Και η Κόζη έχει εγκρίνει την μέθοδο για την σόκτα του Ιουνίου του 11 και του 12. Μετά λοιπόν από αυτά που σας είπα, να σας μιλήσω και για τις δύο συμφωνίες ε, για την διακίνηση ναρκωτικών. Τα πρότεινε η Κόζη στο Συμβούλιο. Η πρώτη συμφωνία αφορά τις διαδρομές κοκαίνης και ηρωίνης. Εγκρίθηκε το 10 υπό την Ισπανική Προεδρία και η δεύτερη αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά ε, που εγκρίθηκε το 12 υπό την Πολωνική Προεδρία. Το πρώτο αφορά τις διαδρομές, όπως σας είπα, κοκαίνης ε, και ηρωίνης αλλά και άλλων μορφών εγκλήματος Υπάρχει ήδη μια τελική έκθεση ε, που αφορά την ανακοπή αυτής της ε, διαδρομής. Ε, αν θέλετε να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε τι είδους προτάσεις έχουν γίνει σχετικά με την εφαρμογή αυτής της έκθεσης. τα προγράμματα αυτά ασχολούνται ε, στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτά ασχολούνται με την ηρωίνη και την κοκαίνη. Πάμε στα συνθετικά ε, ναρκωτικά. Ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για τα συνθετικά ε, ναρκωτικά. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε πλέον χρόνο, για να ολοκληρώσω θέλω να πω βασικά η δική μας η δουλειά είναι η εφαρμογή αυτού του κύκλου πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο για να υπάρχουν προτεραιότητες σε επίπεδο Συμβουλίου. Καλούμεθα να εφαρμόσουμε αυτές τις προτεραιότητες και να συντονίζουμε τις δράσεις στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και κατά ε, του ε, σοβαρού διεθνούς ε, εγκλήματος. Και τελειώνοντας να πω το εξής. Η ΚΟΖΗ εξετάζει και άλλα θέματα που δεν έχουν βέβαια άμεσα σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτικών. Θα αναφέρω μία έκθεση για τη Δυτική Αφρική, πρόσφατα εγκρίθηκε, εκεί γίνεται αξιολόγηση της εφαρμογής των συμπερασμάτων του 2011, ε, την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Ε, η έκθεση αυτή είναι δημοσιευμένη και εκεί μπορείτε να δείτε τα υπέρ και τα κατά των δράσεων στην Δυτική Αφρική. Και θέλω να πω, υπό τη Βολγική Προεδρία ε, οργανώσαμε μια σημαντική ε, εκδήλωση από κοινού με την Interpol ε, για να αξιολογήσουμε την κατάσταση στη Δυτική Αφρική. Και έτσι η Interpol εισήγαγε ένα σύστημα στην Δυτική Αφρική πληροφοριών, το οποίο το χρηματοδοτεί κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Πρόσφατα εξετάσαμε και μία έκθεση της Eurojust. Αυτό, σε αυτό βέβαια θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια, σύντομα. Ε, τέλος, ε, θέλω να φερθώ στην ε, παράνομη διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών. Ε, στη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Υπάρχει και ένα ιταλικό ε, πρόγραμμα για την προστασία της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και με την Κυπριακή Προεδρία εξετάζουμε το πώς μπορούμε όλα αυτά να τα σχετίσουμε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, η Κυπριακή Προεδρία θα πρέπει να ασχοληθεί και με την στρατηγική ε, κατά των ναρκωτικών και κατά της παράνομης διακίνησης ανθρώπινων όντων. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστήκατε και τα 15 λεπτά. Τώρα θα περάσουμε στο γύρο των ερωτήσεων ακούσουμε όλους του συναδέλφους καταρχήν και κατόπιν τις απαντήσεις. Ο ε, κύριος Γεκολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, θα επευθυνθώ στους με τη σειρά. Η ΟΛΑΦ έχει ένα σημαντικό, μια σημαντική δραστηριότητα ελέγχου ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ε, επίσης ε, και στην καταπολεμήση της παραποίησης ακούσαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, αυτή την κοινή επιχείρηση τη ΡΟΚΟ για την καταπολεμήση της λαθρέας εμπορίας τσιγάρων. Έχουμε 10 δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών ε, στον κόσμο από το λαθρομπερίο τσιγάρων. Έτσι λοιπόν ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το θέμα αυτό για να δούμε τι ποιος έχει και στην κατανάλωση των τσιγάρων. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε για ανιχνευσιμότητα των τσιγάρων για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτή τη λαθρέα εμπορία, το λαθρεμπόριο. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν κάποιες βέλτιστες ε, πρακτικές, ε, έγιναν ε, αντικείμενο θέσεις εφαρμογής και υπήρχε μια θετική έκβαση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της καταπολέμησης του οργανωμένου γίνεται λοιπόν, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου η Όλαφ θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ρόλο. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να αναφερθείτε σε αυτό τώρα για την Ευρωπόλ. Ε, αναφερθήκατε στα πλαστά φάρμακα. Πρόκειται για μια αγορά που έχει μεγάλες επιπτώσεις ε, στην υγεία και στην ασφάλεια των πολιτών. Να αναφερθώ όμως ε, στον εκπρόσωπο της Europol. Ε, τι σκέφτεστε για το φάκελο που είναι στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και αφορά την κατάσχεση ε, για να, για να γίνονται πιο αποτελεσματικές κατασχέσεις και σε σχέση με την ΑΚΤΑ, την Εμπορική Συμφωνία κατά τις παραποίησης πρόσφατα. δεν... Ενέκρινε τη συμφωνία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, ε, πώς εντάσσονται αυτά τα στοιχεία και στην οπτική της δικής σας δραστηριότητας. Ε, Κοζή, ε, αναφερθήκατε στα διεθνή εγκλήματα σε οκτώ επιχειρησιακά σχέδια στα Δυτικά Βαλκάνια. Την επόμενη εβδομάδα εμείς ως αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Crime θα επισκεφτούμε τη Σερβία. Εσείς αναφερθήκατε στην ε, αστυνομία, στη συνεργασία με την αστυνομία, στη Σερβία. Πώς λαμβάνει η χώρα αυτή η συνεργασία με την αστυνομία. Εμείς ε, θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα μπορούσαν ε, να υλοποιηθούν και να αναπτυχθούν καλύτερα αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια σε συνεργασία με τη Σερβική Αστυνομία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Newton Down από τους φιλελευθέρους για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για την Όλαφ και τη Europol. Σας ευχαριστούμε που περιγράψατε την επιχείρηση και το ότι βρήκατε στα εμποροκυματοκιβώτια. Βέβαια, ε, όταν ε, δεν υλοποιείται αυτή την επιχείρηση για το υπόλοιπο 99% ε, του έτους, τότε δεν ανοιχνεύουμε τίποτα. Δεν φταίτε εσείς βέβαια, δεν έχετε τους απαραίτητους πόρους για να γίνονται οι έρευνες συνεχώς. Όμως, τι θα μπορούσατε να κάνετε για την Επιτροπή μας, να ζητήσετε τους επικεφαλείς των οργανισμών σας, να μας δώσετε ένα κατάλογο με τις επιθυμίες σας, τι ακριβώς θέλουν οι οργανισμοί την Ευρώπη. Δηλαδή, ποιε αλλαγέ είναι απαραίτητε για να μπορέσετε εσεί ε, να προβαίνετε σε μια συνεχή καταπολέμηση όταν ξεκινήσατε, αναφερθήκατε σε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, που ε, εμποδίζει τις ε, κατασχέσεις κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα μπορούσε αυτή να είναι μία από τις συστάσεις στην εκθεσή σας. Χρειαζόμαστε ένα κατάλογο, ένα shopping list και κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Οτιδήποτε μπορείτε να μας δώσετε προς αυτή την κατεύθυνση σας. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ ήδη γι' αυτό. Τώρα, για τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η παρουσίασή σας. Εγώ ε, επισκέφτηκα και την ιστοσελίδα του ε, Συμβουλίου για να ε, σας ψάξω, όμως ε, τελικά δεν υπάρχεται και δεν βρήκα μία ανακοίνωση τύπου, όμως δεν έλεγε τίποτα, όπως ε, συνήθως. Και πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα, υπάρχει κάποιο μικρό μυστικό μέρος στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, θα μας τα δώσετε εγγράφο. Δυστυχώς, συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά ποιος ε, στην κόζη εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Είναι κάποιος από τη μονίμη αντιπροσωπεία, ο πρεσβευτής ε, ή ε, κάποιος από κάθε πρεσβεία που έρχεται και συμμετέχει στις συζητήσεις. Και πόσοι στη γραμματεία του Συμβουλίου εργάζονται για την κόζη σε σύγκριση με, την, ε, με τους ε, που στέλνουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Νουτοντάν ε, για το ΕΛΚ, η κυρία Ματία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση για τον εκπρόσωπο της Όλαφ. Θα ήθελα να μου πείτε ε, ποια είναι τα προϊόντα της κατάσχεσης για τον κύριο της Γεροπόλ, δεν ξέρω. Όταν ε, έχουμε κάποια αγαθά που κατάσχεται, δηλαδή ακούσαμε χιλιάδες τόνους τσιγάρων, ε, είναι εντυπωσιακό κάτι τέτοιο. Τι συμβαίνει συγκεκριμένα, πού ε, πάνε αυτά τα προϊόντα, πού τα βάζετε και όταν έχουμε κοινέ επιχειρήσεις όπου συμμετέχουν πολλά κρατημέλη, πώς υλοποιούνται, πώς γίνεται η κατανομή. Θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα πώ υλοποιείται αυτή η επιχείρηση όταν είστε σε ένα λιμάνι, παραδείγματο χάρη. Τι ακριβώ κάνετε. Και σε σχέση και όσα ρώτησε ο συνάδελφος Νιτοντάν. Δεν έχουμε ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τις απώλειες ε, σε επίπεδο ΦΠΑ παραδείγματος χάρη ένα κράτος μέλος ότι έχουμε τόσες απώλειες ε, από τα έσοδα του ΦΠΑ ή ανά επιχείρηση γιατί το εμπορίο τσιγάρων παραδείγματος χάρη να λέμε ότι για τη μου σημαίνει τόση απώλεια εσόδων. Δηλαδή ε, θέλουμε τα στοιχεία για να ξέρουμε ότι παίρνουμε το χάρη για ε, τις επιχειρήσεις, τις αυτό σημαίνει τόσο για την αυτοβιομηχανία. Ε, έχουμε αυτά τα νούμερα γιατί παίρνει το χάρη. Ακόμη και αν ε, πάει κανείς ε, σε ένα γκαράζ μπορεί να του δώσουν και ένα ανταλλακτικό παραποιημένο. Και μιλήσατε και για τα παρασιτοκτόνα και αυτό είναι απίστευτο. Πρώτη φορά άκουσα εγώ να γίνεται λόγος γι' αυτό σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Εδώ μας κάνετε να ανακαλύπτουμε κάτι. Όμως ε, από ό,τι φαίνεται περνάει από ένα επαγγελματικό κύκλωμα. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, έχουμε τους ε, γεωργούς που πάνε να ψάξουν τι πρέπει να θα βάλουν στον κήπο τους. Έχουμε δηλαδή αρκετά εύκολη διέλευση από επαγγελματικά κυκλώματα, όμως νομίζω ότι θα μπορούσε να σταματήσει κάτι τέτοιο, γιατί φαντάζομαι ότι μεγάλη γεωργοί τελικά περνούν από εσωτερικά δίκτυα επαγγελματικά για να προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα και πραγματικά εμένα με εντυπωσιάσει αυτό. Αυτό ζημιώνει πάρα πολύ το περιβάλλον. Δεν κατανοώ λοιπόν πώς μπορεί να είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Και κυρίως να υπάρχει αύξηση κατανάλωσης, τεράστια κατανάλωση λιπασμάτων, ε, παρασιτοκτόνων. Και ήθελα να θέσω την ερώτηση, καθώ έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπο τη Κόζη. Η Γεροπόλη έχει πραγματικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει και αύξηση τη εμπιστοσύνη των κρατών μελών για να συμμετέχουν σε επιχειρησιακό επίπεδο και λειτουργούν τα πράγματα, γιατί μερικές φορές ε, ξέρουμε ότι είναι ακριβώς διστακτικά τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν μαζί σε τέτοιες επιχειρήσεις Και ε, θα πρέπει να πείσετε ορισμένα. Χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ η Κόζη για να μα πει σε ποιο βαθμό συνεχίζεται να αυξάνεται αυτή η εμπιστοσύνη από την πλευρά των κρατών μελών. Και μια τελευταία ερώτηση για τα αραβικά μοιράτα και θα σταματήσω. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε προσφέρει βιομηχανία στην ΟΕΕ Μοιράτα για το οργανωμένο έγκλημα και θα ήθελα να μου πείτε γιατί ε, σημειώνεται αυτή η αύξηση στα παραπημένα αγαθά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κυλακάκης, παρακαλώ. Thank you and first of all, thank Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Έχω τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις ε, σε σχέση με τα παραπημένα αγαθά και την παράνομη διακίνηση. Τρεις μάλλον ερωτήσεις. Καταρχήν, ποια είναι τα έσοδα που χάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών, ποια είναι τα πολλαστατά έσοδα από αυτέ τι δραστηριότητε, Έχετε κάποια ιδέα για το μέγεθο. Και ποιοι είναι οι πόροι που χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των δύο αυτών προβλημάτων. Έχουμε πρόβλημα πόρων, κατά την άποψή σα. Δηλαδή δεν έχουμε επαρκή πόρους. Σε σχέση με τα έσοδα που χάνουμε ιδίω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι το θέμα της πεκορικότητας. Βλέπετε να υπάρχει ανάγκη αύξησης πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί αν αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε επίπεδο κρατών μελών. Η δεύτερη ερώτησή μου σχετίζεται με τη διαφθορά. Η εκπρόσωπος του UNODC είπε ότι υπάρχουν ε, διαδρομές διαφθοράς παράλληλες με τις οδούς διακίνησης ναρκωτικών. Και υποθέτω ότι οι ίδιες οδοί που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των ναρκωτικών, οι ίδιες οδοί διαφθοράς χρησιμοποιούνται και για την παραποίηση για άλλες δραστηριότητες, γιατί ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος δέχεται να δωροδοκηθεί για κάτι, θα δεχτεί να δωροδοκηθεί και για άλλα αγαθά. οι οργανισμοί σας έχουν εντοπίσει αυτές τις οδούς διαφθοράς. Γιατί μια στρατηγική είναι η καταπολέμηση για να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τους εγκληματίες, όμως μια διαφορετική στρατηγική είναι να συλληφθούν όσοι διευκολύνουν τη δουλειά των εγκληματιών. Έχετε εργαστεί λοιπόν από αυτού Και ιδίω αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και όμορες χώρες με τι οποίε έχουμε πολύ καλές σχέσεις και δεπανούμε χρήματα. Και ένας μεγάλος βαθμό ε, αυτή της διαφοράς παρατηρείται σε αυτές τις όμορες χώρες. Έτσι λοιπόν υποθέτω, αν ε, εμπορία ανθρώπων περνά ε, από κάποια σύνορα, αν πάμε στους αξιωματούχους στη γειτονική μας χώρα εκεί και θέσουμε το θέμα της διαφθοράς, θα δούμε ότι υπάρχει εκεί ένας μεγάλος αριθμός του προσωπικού που δωροδοκείται. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτές τις ε, διαδρομές διαφθοράς, πώς μπορούμε να τις, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο πιο δύναμος κρίκος της και Κάτι Υπάρχουν πολλά χρήματα που προέρχονται στον ευρωπαϊκό προβλησμό από τι καπνοβιομηχανίε. για την καταπολέμηση των ε, παραπημένων τσιγάρων. Νομίζω ότι μιλάμε για ένα ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Θέλω να ρωτήσω, πού πάνε αυτά τα χρήματα, ποιος τα δαπανά και ποια είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω να κάνω μόνο κάποιες ε, σύντομες ερωτήσεις ε, που θα συμπληρώσουν αυτά τα οποία ρώτησαν οι συνάδελφοι. Και η πρώτη μου λιγάκι ε, προκλητική ερώτηση είναι το εξής. Λέτε ότι η συνεργασία είναι το σημαντικότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι πάει πάρα πολύ καλά. Με τις ε, τρεις εισηγήσεις που άκουσα ε, κατέληξα στο ότι υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις. Ίσως ε, λοιπόν πολλοί πόροι να χρησιμοποιούνται απλά και μόνο στο συντονισμό. Μήπως εντωμεταξύ έχουμε πολλούς περισσότερους από ό,τι πρέπει οργανισμούς. Όχι λιγότερους, αλλά περισσότερους. Γιατί η συνεργασία είναι σημαντική και πρέπει να μας το ξεκαθαρίζετε. Από το Συμβούλιο ακούστηκε ότι ορισμένα κρατημέλη που έχουν βέβαια πόρους είναι αρμόδια για ορισμένου τομεί εγκλήματο. Ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε, κυρίως ας πούμε, τι κάνει η Γερμανία και ποια είναι η χώρα που ασχολείται ιδιαίτερα με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, ίσως να το ξέρετε. Ε, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου αφορά αυτό που είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε ακόμα, οι οδηγίες που έχουμε αρκούν για σας, γιατί έχουμε οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε επίσης ε, ένα νόμο ε, για την αντιμετώπιση των παραποιημένων φαρμάκων. Στην αρμόδια επιτροπή επικρίναμε το ότι η οδηγία αυτή δεν περιλαμβάνει τις online πωλήσει παρά μόνο τις υπόλοιπες. Ε, επίσης, θα θέλαμε να μας πείτε κατά την άποψη σας πού υπάρχουν ελλείμματα στο νομικό τομέα. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί αν πράγματι ισχύει αυτό που είπατε, ότι δεν είναι δυνατόν να κατάσχονται ε, προϊόντα που βρίσκονται σε διαμετακόμιση, αυτό είναι φοβερό. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο στις ε, συμφωνίες FTA να ε, λαμβάνονται μέτρα για χώρες οι οποίες ε, εισάγουν προϊόντα σε εμά, γιατί αυτές οι συμφωνίες, η FTA, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Τέλος, είπατε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους στα διάφορα προϊόντα. Ε, όσον αφορά τα παραποιημένα φάρμακα, μου είναι αυτονόητο και για τα πολυτελή αγαθά. Όμως ε, υπάρχουν και πολλά ε, πάμφτινα προϊόντα, ας πούμε τα τσιγάρα. Εκεί δεν παίζει ρόλο το ίδιο το προϊόν, αλλά η ποσότητα, ο όγκος. Ίσως λοιπόν μπορείτε να μας εξηγήσετε πού ακριβώ είναι μεγάλο το περιθώριο κέρδους. Και τέλος να πω ότι όσον αφορά τη Γερμανία, ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία, τι κάνουν τα προϊόντα που κατάσχονται. Ας πούμε στη Γερμανία Ξέρω ότι όταν τα τελωνία κατάσχουν προϊόντα καταστρέφονται εκείνη τη στιγμή και παντελώς για να μην ξαναμπούν στην αλυσίδα. Δεν ξέρω όμως αν το κάνουν αυτό όλες οι χώρες. Πάρα πολύ ωραία. Σόνταγκαρτ παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να μην κατάλαβα καλά να μιλήσουμε για τα αντίγραφα και για προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο όγκος της παραποίησης και των περιοτικών προϊόντων που παράγονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που εξάγονται από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Παραδείγματος χάρη δεν μιλάμε για φάρμακα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Όταν μιλάμε για προστοκτόνα, είναι σαφές ότι μιλάμε για ένα μεγάλο πρόβλημα όταν μιλάμε για παραπημένα προϊόντα, αλλά υπάρχει και το εξή στοιχείο ότι έχουμε μια δυσκολία ότι διαφέρει η νομοθεσία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα παραστοκτόνα. Υπάρχουν λοιπόν νόμιμα παραστοκτόνα που κυκλοφορούν, που διακινούνται σε άλλε χώρε ή μιλάμε για προϊόντα απαγορευμένα. Μία σειρά παραδείγματο χάρη που μπορεί να επιτρέπεται στην Πολωνία και να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία του σε άλλε χώρε, όπω στη Σουηδία, στη Δανία. Στο πλαίσιο των ερευνών σα αντιμετωπίσατε συναντήσατε τέτοια προϊόντα νόμιμα που όμως είναι αντικείμενο διακίνησης. Ευχαριστώ κύριε Σόντεργκατ Πριν να ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλεισμένους μας, ε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αν ε, και οι ερωτήσει των συναδέλφων ήταν αρκετά σαφείς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πτυχή που ανέφερε ο κύριος Σκυλακάκης. Ε, αναφερθήκε στη διαφθορά. Αν όλα αυτά είναι δυνατά, μας το είπε και πριν η κυρία Με, αν όλα αυτά είναι δυνατά και σε επίπεδο παραποίηση. Ε, προφανώς αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα καλά παγιωμένο κύκλωμα και έχουμε δει αρκετά υψηλά αριθμητικά στοιχεία. Μιλάμε για πηγές που έχουν επίπτωση στην υγεία των καταναλωτών, σημαντική επίπτωση. Αν λοιπόν όλα αυτά ήταν δυνατά και συνεχίζουν να είναι δυνατά, προφανώς σε αυτό το τομέα, στον αποκαλέσουμε έτσι, η διαφθορά συνεχίζει να έχει ένα μεγάλο περιθώριο. Ε, και μιλάμε και για τους στελωνιακούς, αλλά και για άτομα που στελεχώνουν διάφορους θεσμούς, διάφορους φορούς και σε κάποιο σημείο αυτού του κυκλώματος καθώς αποτελούν τμήμα αυτού επιτρέπουν με τη βούλησή τους ε, την διεύρυνση αυτής της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία Θα κάνω μία ερώτηση που ίσως να σας φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά για μας είναι σημαντικό να καταλάβουμε. Τα κράτη-μέλη πόσο επενδύουν στην πραγματικότητα και πόσο πιστεύουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Εγώ πολλές φορές έχω συνομιλήσει με τον διευθυντή της Europol, τον κ. Ράιτ και μαζί, ε, έχουμε δηλώσει την αναγκαιότητα τα κράτη-μέλη να πιστέψουν πραγματικά σε αυτούς τους οργανισμούς για να μπορεί να γίνει αυτό το παιδικό άλμα. και προλίγου είδαμε πραγματικά τεράστιες ποσότητες ε, φαρμάκων και παραστοκτώνων που έχουν κατασχεθεί και αφού κατασχεθούν ε, καταστρέφονται φυσικά τα προϊόντα αυτά γιατί δεν μπορούν ε, να ξανατεθούν, για να μην ξανατεθούν πλέον εκ νέου σε μια αγορά παράνομη. Το κύριο όγκο αυτών φτάνει από την Κίνα. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ουσιαστικά ε, τηρεί και θέτει σε εφαρμογή την συμβατική της ικανότητα σε αυτό το τομέα και αυτό δεν το ρωτώ μόνο για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Κίνα γιατί ξέρετε ότι είναι αντικείμενο εκμετάλλευση από ένα τέτοιο κύκλωμα. Όλα αυτά, όπως ρώτησαν ε, ήδη συνάδελφοι. βρίσκει μια πολιτική ικανοποιητική δράση από την πλευρά του Κοινοβουλίου, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πιστεύετε από νομοθετική σκοπιά, από επιχειρησιακή σκοπιά, να αυξήσουμε κατά κάποιο τρόπο όλα όσα κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια ακόμη πιο συγκεκριμένη συνεργασία. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Ένα και κατόπιν ε, στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο καθένας ε, έχει πέντε λεπτά για να απαντήσει. Καταρχήν ο κύριο Ένα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ένα από τα κυρία καθήκοντα της Όλαφ ε, είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων, αλλά πέραν αυτού του καθήκοντος έχουμε και το καθήκον της καταπολέμησης της παραποίησης. Ε, και είναι αλήθεια ότι τα τσιγάρα εντάσσονται σε αυτό το τομέα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωση, Ό,τι αφορά άλλου είδους αγαθά, εδώ έχουμε αντίκτυπο σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο δημόσια υγεία αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, αν αυτά είναι διαφορετικά, αλλά και οι δύο συνιστώσει είναι σημαντικέ ε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του Ντζον για ε, τον κατάλογο των επιθυμιών. Βεβαίω, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ τη διευκόλυνση του εμπορίου, γιατί θέλουμε τη διευκόλυνση του εμπορίου και αφετέρου τη διαχείριση του κινδύνου και πρέπει να βρούμε και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε το λαθρεμπόριο. Μία από τις λύσεις ε, που έχουμε σκεφτεί σε επίπεδο κομισιών είναι ακριβώς να δώσουμε έμφαση ε, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές σε άμεσες κινήσεις. Τώρα η Όλαφ έχει ε, πρόσβαση για τη διαμετακόμιση, αλλά όχι για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Αυτό θα ήταν σημαντική πρόοδος. Αναφερθήκατε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Βεβαίως η απόφαση αυτή για τη διαμετακόμιση μας ανησυχεί, οι υπηρεσίε τη Κομισιόν εργάζονται για την εξέβρεση πιο οριστική λύση, αλλά εν τω μεταξύ ο ΛΑΦ προτείνει μια ρεαλιστική λύση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ε, οι συμφωνίε αμοιβαία συνδρομή με τι τρίτε χώρε για να ενημερώνονται συστηματικά οι τρίτε χώρε για το κίνδυνο παραποίηση. Και αυτό που κάναμε μέχρι τώρα ε, με την Αίγυπτο, αυτό ήταν όταν είχαμε αυτή την έρευνα για τα φάρμακα και η Αίγυπτος μα στέλνει πληροφορίε σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Αναφέρατε το γεγονό ότι ε, μπορεί να υπάρχει και κάποια δωροδοκία στον, στον ε, τομέα του τελωνία. Τώρα, ε, οι υπηρεσίες καταθέτουν τις πληροφορίες. Δεν χρειάζεται ο εισαγωγής ή ο να κάνει τη διασάφηση. Αυτό ε, πρέπει να το δούμε για τη διαχείριση του κινδύνου και για την καταπολέμηση της παραποίησης. Η κυρία Ματιέ μας ρώτησε τι γίνεται με τα εμπορεύματα αυτά, αφού τα εμπορεύματα ε, κρατούνται στο τελωνείο τίθεται σε ένα καθεστώς ανασταλτικός προς τους δασμούς και ε, ο κάτοχος ε, του εμπορεύματο πρέπει να πληρώσει τις δαπάνες της αποθήκευσης μέχρι να υπάρχει κάποια απόφαση του δικαστηρίου για την καταστροφή ή για την επίδοση. Ε, και αφού υπάρχει καταστροφή, αν υπάρξει καταστροφή μπορεί ο κάτοχος να στραφεί στο αυτόν που το προμήθευσε για να αποζημωθεί Πρόκειται για υποχρέωση λοιπόν καταστροφής των εμπορευμάτων, όλα τα τελωνία έτσι λειτουργούν. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόβλημα των πόρων. Χρειαζόμαστε όσο δυνατόν μεγαλύτερη καινοτομία και νομίζω ότι η καινοτομία περνά και από τις βάσεις δεδομένων που θα πρέπει να εμπλουτιστούν το δυνατόν περισσότερο και αν μπορούμε να αντιλάσσουμε τις πληροφορίες. σημείωσα ότι δεν υπάρχει καμία επικάλυψη μεταξύ δραστηριών Όλαφ και Γιουροπόλ. σε ό,τι αφορά την παραποίηση. Ο Όλαφ έχει διοικητικέ αρμοδιότητε έρευνα. Δεν μπορούμε να λάβουμε δράση στον ποινικό τομέα, ενώ η Γιουροπόλ έχει αρμοδιότητε που δεν καλύπτει τη διοικητική έρευνα. Εμεί ε, μπορούμε να συλλέξουμε αποδείξει που χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια και 150 τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα ασκήσουν τι διώξει. Η αρμοδιότητα κατά συνάδελφους ε, έχουν να κάνουν ε, με το οργανωμένο έγκλημα περισσότερο. Πραγματικά είμαστε ανάντι του σταδίου αυτού και η συνεργασία μεταξύ του διοικητικού και του ποινικού τομέα είναι σημαντική γιατί τότε μπορούμε ακριβώς να αξιολογήσουμε ε, το μέγεθος της απάτης. Δεν έχουμε φυσικά αριθμητικά στοιχεία ε, για την ιστορική αγορά και γι' αυτό ε, ιδρύσαμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραποίηση που βρίσκεται στο Αλικάντα και θα αξιολογήσει την κατάσταση σε επίπεδο ιστορική αγοράς. Σε επίπεδο τελωνίων έχουμε ένα μηχανισμό που το διαχειρίζεται η ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΤΑΞΟΥΝΤ και στο πλαίσιο του κανονισμού 1383-2003 έχουμε ένα μηχανισμό στατιστικών. Στο μελλοντικό κανονισμό που είναι διαπραγμάτευση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα είναι η κυρία Κρότσμαν. Λέμε ότι τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να εισάγουν δύο ή τρεις φορές τις ίδιες πληροφορίες γιατί συχνά ζητούνται οι ίδιες πληροφορίες στις ελληνικές αρχές. Ξέβρεμε ένα μηχανισμό και θα δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την συνεργασία και την μοναδική καταχώρηση των πληροφοριών και θα μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και ελπίζουμε να δίνονται αυτές ε, οι πληροφορίες στη Europol και θα υπάρχουν και ονόματα εκεί, ενώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων θα γίνονται χωρίς ονόματα. Στη συνέχεια σημείωσα και το πρόβλημα των εμπορικών ε, συμφωνιών για την ΕΣΕΣ. Και στο πλαίσιο του ΣΕΑΝ έχουμε δράσεις με τη τελωνία των ασιατικών χωρών, έχουμε τις επιχειρήσεις Διάμπολο 1 και 2 με τη συνεργασία της Ιντερπόλ και εκεί ε, λάβαμε εντολή για να συνεχίσουμε αυτή τη δράση και συμμετείχαν 19 σχετικές χώρες Έχουμε 50 ε, χώρε που εκπροσωπούν τι Ευρωπαϊκέ Ένωση και τι χώρε τη Ασία και αυτέ οι 50 χώρε έχουν αποφασίσει να υλοποιήσουν συγκεκριμένε δράσει. Και ελπίζουμε τώρα ότι θα υπάρξει νέα ανάληψη πρωτοβουλία από τι ε, κινέζικε αρχέ. Γιατί τα κινέζικα τελωνία δεν έχουν διοικητικέ αρμοδιότητε και αυτό μα θέτει πρόβλημα. Αντίθετα, η κινέζικη αστυνομία έχει αποφασίσει να δράσει και θα πρέπει στην Κοινή Επιτροπή με την Κίνα να προσπαθήσουμε να φέρουμε την ε, αστυνομία της Κίνας ως αρμόδια αρχή με τέτοια καθήκοντα που έχουν και οι υπόλοιπες αρχές έτσι ώστε θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε επίπεδο διοικητικής έρευνας και νομίζω τώρα δεν μπορώ να δώσω το λόγο στους αδέλφους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαστερκίστη. Ε, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τα προϊόντα τα οποία έρχονται και κατέσχονται ως πλαστά ή από λαθρεμπόριο. Εμείς προσπαθούμε, προσωπικά τουλάχιστον πιστεύω ότι έξι μήνες, ένα χρόνο μπορεί να βρεθεί κάποιος στη φυλακή, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα κέρδη. Ο πιο αποτελεσματικό τρόπος είναι να ξέρει ο εγκληματίας ότι δεν πρόκειται να δοποδοθούν ποτέ τα προϊόντα αυτά. Έχουμε λοιπόν συνεργασία σε αυτό και με την Ισπανία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την ΕΚΑ που είναι η υπηρεσία ε, η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό της ε, Επίδοση των ε, προϊόντων ε, εγκληματικής πράξης. Εννοείται ότι τα πλαστά, ε, φάρμακα για παράδειγμα, δεν επιστρέφονται. Για να έρθω τώρα στην ερώτηση του κυρίου Νιούτον. Πιστεύω ότι μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες μας είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι στην δικαιοσύνη ε, ή στην κοινή γνώμη δεν αντιλαμβάνονται. Δεν, τους, δεν ευαισθητοποιούνται για το θέμα των, των πλαστών προϊόντων. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πίσω από αυτά τα πλαστά προϊόντα υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις που δρούν εντελώς επαγγελματικά, χωρίς κανένα δισταγμό να βάλουν πλαστά προϊόντα στην αγορά, τα οποία μπορεί να είναι ακόμα και επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Όσον αφορά τη συνεργασία τώρα με τις χώρες μέλη, μέχρι τώρα πηγαίνει πολύ καλά από πλευρά της Europol. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο καλύτερος ε, τρόπος να γίνει γνωστή η δουλειά μας είναι από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, όταν υπάρξει μια επιχείρηση η οποία πάει καλά, αυτό το μαθαίνει ο κόσμος όσον αφορά τα νούμερα και τη τάση τους. Κοιτάξτε, η στατιστική μας είναι όντως ένα δύναμο σημείο. Για τα πλαστά προϊόντα και για την πειρατεία υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη. Ο ΣΑΚΑ έκανε μια μελέτη, όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 200 με 250 δισεκατομμύρια δολάρια απώλεια εκτίμησε ότι έχουμε. εξαιτία του το πλαστό επίση εμπόριο είναι κάπου 3 με 3,5% στο διεθνές εμπόριο. Αλλά δυστυχώ δεν έχω τίποτα πιο συγκεκριμένο. Ρωτήσατε αν θέλουμε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό ή μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις εγκληματικές δραστηριότητες γύρω από τα πλαστά ε, προϊόντα και την πειρατεία. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο σε καθημερινή βάση ασχολούνται με τα πλαστά και την παραπίση και άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι εγκληματικέ οργανώσεις ασχολούνται όλο και περισσότερο με τα πλαστά προϊόντα γιατί διαπιστώνουν ε, προφανώς ότι τους αποφέρουν περισσότερα. Σιγαρέτα επίσης είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε κάποιο προπολογισμό, το χρησιμοποιούμε βέβαια. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω γι' αυτό τίποτα περισσότερο. Για την επικάλυψη τώρα των διαφόρων ε, μονάδων. Μα, ε, εντάξει, συνεργαζόμαστε, δουλεύουμε για το θέμα των πλαστών ε, μαζί η Όλαφ και εμείς. Μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι επικάλυψη. Η Europol και η Interpol επίσης συνεργάζονται όσον αφορά τα πλαστά τρόφιμα και ποτά. αλλά η Europol ασχολείται περισσότερο με τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Interpol με τις υπόλοιπες χώρες. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει συνεργασία για να αποφευθεί η επικάλυψη. Εξάλλου το είπε και ο συνάδελφος Μουτχερή, όταν πρόκειται για διοικητικές διαδικασίες, ασχολούμαστε ο καθένας με κάποιες ε, οργανώσεις. Τα τελωνία περισσότερο με τα αγαθά, ε, άλλοι περισσότερο με τις εγκληματικές οργανώσεις. Οπότε, ένα θέμα είναι η κατάσχεση προϊόντος. Από εκεί και πέρα, το να φτάσουμε στους πραγματικούς εγκληματίες, που δεν φτάνουμε πάντα με επιτυχία, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει, να φτάσουμε στους εγκληματίες. Τέλος, για την παραγωγή της επιπτώσεις της παραγωγής της Κίνας, αυτό που ξέχασα να σας πω στην παρουσίασή μου αρχικά είναι ότι υπάρχει μια νέα τάση, ότι δηλαδή η τελική παραγωγή όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται σε μας. Ότι δηλαδή μπαίνουν κοντέινερ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλαστά, πόλος ή μπλουζάκια κτλ. Οι ετικέτες όμως μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι έγινε μια κατάσχεση στη Χάγη από την Ολλανδική Υπηρεσία, 2 χιλιόμετρα από την Europol δηλαδή, με πλαστά προϊόντα. Για να σας δώσω δηλαδή ένα παράδειγμα και στο Παρίσι, στο Βελιέ για παράδειγμα, επίσης ήταν καμιά δεκαριά που πήγαν από τη Χάγη μέσω Αμβέρσα στο Τεβελιέ και εκεί πήγανε τίσερτ χωρί χωρίς ετικέτες για να μπουν ετικέτες. Άρα είναι πράγματα που γίνονται και στις χώρες μας. Αυτό ήθελα ακόμα να προσθέσω, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τελευταία παρέμβαση τώρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό που ρώτησε ο κ. Γιακολίνο για τη Σερβία. Καλύπτεται από το σχέδιό μας για τα Δυτικά Βαλκάνια και είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την Ιταλία. Η Ιταλία είναι προτερότητά μας. Γιατί έχουμε εγκληματική δραστηριότητα από αυτή την περιοχή. Τώρα σε επίπεδο Europol έχουμε πάρα πολλέ ε, συνεδριάσεις που κάνουμε για να καλύψουμε όλες τις χώρες οι οποίες σε θελοντική βάση συμμετέχουν στην επιχειρησιακή δράση. Τώρα η δράση αυτή καθε αυτή επιτόπου βασίζεται στι διμερεί δράσει των χωρών μελών. Οι χώρε δηλαδή είναι εκείνε, οι οποίε προχωρούν σε περισσιακέ δράσει για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδου εγκληματικότητα. Και μπορούμε να προβλέψουμε βέβαια και τη συμμετοχή των αξιωματούχων σύνδεση που βρίσκονται επί τόπου. Αυτό που δεν έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, είναι διαρθρωμένο διάλογο με τη Σερβία για το κόζι. Δεν έχουμε τέτοιο διάλογο για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Σερβία στα πλαίσια του Κόζη. Στα πλαίσια των δράσεων και διμερός υπάρχει συνεργασία. Για την ερώτηση του κύριου Νιούτον Ντάν για τα απόρριτα έγγραφα. Όντω, μερικέ φορέ είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε όλα τα έγγραφα του Συμβουλίου να βρει κανεί ε, ό,τι έχει να κάνει με το κόζι. Πάντως υπάρχουν ε, στη Standard Committee αναφορές για τα διάβαρα έγγραφα που έχουν να κάνουν με αυτά. Υπάρχουν αριθμοί αναφοράς για το κάθε έγγραφο. Δεν είναι όλα δημόσια φυσικά, αλλά υπάρχουν στο Συμβούλιο. Εννοείται ότι πρέπει να δουλέψετε με τους αριθμούς αναφοράς για να προχωρήσετε. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για το κόσι Είναι μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Και ισχύει για την διαφάνεια ότι ισχύει και για όλα τα έγγραφα του Συμβουλίου. Τώρα για την εκπροσώπηση των κρατών μελών ε, στη ΚΟΣΗ. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Δεν είναι απόφαση του Συμβουλίου, δεν αποφασίζει το Συμβούλιο ποια αντιπροσωπή θα στείλει το κάθε κράτο μέλο. Ε, βασίζονται στι Βρυξέλλε. Οι περισσότεροι έρχονται λοιπόν από τι πρωτεύουσε. Ορισμένε χώρε θέλουν του επικεφαλεί των ε, αστυνομιών του, στο Βέλγιο ή η Ισπανία για παράδειγμα. Είναι ο κομισέραν σεφ. Άλλοι στέλνουν ε, υψηλού αξιωματούχου του Υπουργείου Δικαιοσύνη ή Εσωτερικών, Σουηδία και Γερμανία. Και κάποιοι λίγοι στέλνουν συναδέλφους από τη μόνιμη αντιπροσωπεία, η Σλοβενία για παράδειγμα. Οι περισσότεροι πάντως έρχονται από τις πρωτεύουσες και είναι είτε από την αστυνομία είτε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνη. Τώρα για την Γενική Γραμματεία έχουμε μια μικρή ομάδα που δουλεύει για την κόζη. Έχουμε πολιτικητικούς, έχουμε δύο εθνικούς επιρρογνώμονες και δύο βοηθούς που συμπληρώνουν τη δουλειά της κόζη. Για να απαντήσω στην κυρία Ματιέ. Αναφέρθηκα λίγο στο θέμα της εμπιστευτικότητας. Υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις χώρες μέλη για να συνεργαστούν. Για την αστυνομική συνεργασία νομίζω ότι δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα πόρων. Οι υπηρεσίες της αστυνομίας που είναι αρμόδιες για την εσωτερική ασφάλεια έχουν να αντιμετωπίσουν και τα εσωτερικά προβλήματα. Άρα μένουν ελάχιστοι πόροι για να αφιερωθούν στις ευρωπαϊκές δράσεις. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, να βρεθούν επιπλέον πόροι δηλαδή για να φτάσουν και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια σχέδια. Αυτό που ρωτάτε συνέχεια είναι για τη χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, πολλές χώρες θα θέλανε τα ευρωπαϊκά σχέδια να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να την έχουμε. Το είδαμε και με τις μικτές ερευνητικέ ομάδες. Η Eurojust είχε έναν προπολογισμό για αυτές τις κοινέ ομάδες, τον προπολογισμό, αλλά ο προπολογισμό αυτός θα εξαφανιστεί όπου να είναι. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε πολλές χώρες μέλη, να μην μπορούμε δηλαδή πια από κοινού να χρηματοδοτούμε τέτοιες έρευνες. Οπότε περισσότερο από θέμα εμπιστοσύνη θα έλεγα ότι είναι θέμα χρηματοδότησης και πόρων για το θέμα των επικαλύψεων. όπω και οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελάχιστη επικάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διάφοροι, τα διάφορα όργανα έχουν το δικό του τομέα δράση, μπορεί να ασχολούνται με το ίδιο θέμα, οργανωμένο έγκλημα για παράδειγμα, αλλά τα μέσα δράσης που διαθέτουν είναι διαφορετικά. Η Eurojust, η Europol, η Frontex, η Olaf έχουν διαφορετικά μέσα δράση αλλά τον ίδιο στόχο, άρα δεν υπάρχει επικάλυψη. Κίνδυνο επικάλυψη υπάρχει όταν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Europol δηλαδή να κάνει τέτοια πράγματα που κάνει και η Interpol εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έχουμε μηχανισμού διαλόγου, συζητήσεων μεταξύ μα. και όταν βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Interpol έχει ήδη ένα σχέδιο, μια δράση που ανταποκρίνεται στι δικέ μα ανάγκε, δεν θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και εμεί στην Ευρώπη. Θα δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε από την Interpol. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί όπω είναι το COSI, ώστε να προκύπτει ο συντονισμό αυτό για να μην υπάρχουν ούτε επικαλύψει, αλλά ούτε και κενά στη συνεργασία μα. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή των κρατών μελών στι διάφορε επιχειρησιακέ δράσει είναι σε θελοντική βάση. Τα κράτη δεν είναι υποχρεωμένα όλα να συμμετέχουν στι δράσει αυτέ, συμμετέχουν σε θελοντική βάση όπω είπα. Για τη Γερμανία, για παράδειγμα, η Γερμανία συμμετέχει πολύ στα Δυτικά Βαλκάνια για την εμπορία ανθρώπων ή ηρωίνη. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Έχουν ζητήσει το λόγο και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ξεκινάμε με τον συνάδελφο Νιούτον Ντάν. Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που είπε ο συνάδελφος, ο κύριος από τη Europol. Είπε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι το να υπάρξει ευαισθητοποίηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ουσία των πάντων. Διότι αν μπορούμε να επιτύχουμε την ε, συνειδητοποίηση του κοινού ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, θα βοηθήσουν και θα πούνε επίσης «Μα κάνετε και κάτι». Και έτσι θα προκύψει πολιτική δράση, διότι οι πολιτικοί ε, τείνουν να αντιδρούν στην ε, δράση. Πώς λοιπόν θα υπάρξει ευαισθητοποίηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη συζήτηση που είχα με τον πρώτο διευθυντή της Europol, ένα θαυμάσιο Γερμανό που μετά επέστρεψε στο Βερολίνο. Πώς μπορεί να υπάρξει ευαισθητοποίηση και είπε, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι η 11η Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη. Αυτή η τεράστια επίθεση από το οργανωμένο έγκλημα, όπου όλοι στην Ευρώπη έλεγαν γιατί έγινε αυτό ε, και τι πρέπει να κάνετε. Ε, Βεβαίω, είπε δεν πρέπει να καταλήγουμε εκεί. Αυτή δεν είναι η λύση. Η λύση λοιπόν που εγώ προτείνω είναι η Επιτροπή αυτή ε, και οι συζητήσεις ε, που θα έχουμε στην Ολομέλεια αυτά να αποτελούν ε, ένα σημαντικό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οτιδήποτε λοιπόν μπορείτε να μας προσφέρετε για την ευαισθητοποίηση θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι η έκκλησή μου. Και θέλω και άλλη μια ερώτηση. Για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, τι θα λέγατε ε, να αναφερθούν στην ισοσυλία της ε, Europol οι 10 καταζητούμενοι ε, οι πιο σκληροί καταζητούμενοι. Να έχουμε τους 10 σκληρούς ε, καταζητούμενους στην Ευρώπη από τη Europol, όπως συμβαίνει στη συστοθελίδες του FBI. Ε, και αυτό νομίζω θα βοηθούσε στο να υπάρχει καλύτερη ευαισθητοποίηση. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Βάιλερ έχει το λόγο. Η κυρία Βάιλερ. Η κυρία Μπάιλερ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επειδή έχουμε αρκετό χρόνο, θέλω και εγώ να κάνω μία ερώτηση. Καταρχήν, όσον αφορά αυτά που λέγησαν προηγουμένως, ε, κοιτάξτε, έχουμε έναν πολύ καλό σύμμαχο, τα μέσα ενημέρωσης. Πριν από δύο εβδομάδες ε, διαβάσαμε ένα ε, μεγάλο άρθρο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ε, για την Όλαφ, για τις απάτες. Τα μέσα ενημέρωσης τα βγάζουν αυτά προς τα έξω. Σε εμά στη Γερμανία τα παραποιημένα φάρμακα είναι ένα τεράστιο θέμα οποτεδήποτε ε, συλλαμβάνουν κάποιον. Έχουμε εδώ τους ε, καλύτερους ε, συμμάχους. Επίσης, να πω ότι έχουμε και την υποστήριξη της κοινή γνώμης. Οι ομάδες Δίωξη του εγκλήματος ε, είναι σωστά εξοπλισμένες. Εγώ λοιπόν δεν έχω ακούσει αρνητική κριτική γιατί κατά τα άλλα πολύ εύκολα ασκείται κριτική κατά της Ευρώπης. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει και υποστήριξη της κοινή γνώμης. Θα ήθελα να ακούσω λιγάκι και τι γίνεται με τα τελωνία. Εγώ κανονικά είμαι στην Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς ε, και εκεί έχουμε μεταρρύθμιση, αποφασίσαμε για τη μεταρρύθμιση του τελωνιακού κώδικα και η βιομηχανία ε, διαφωνεί ριζικά. Τουλάχιστον η γερμανική, η βρετανική και η γαλλική ε, βιομηχανία. Και ρωτώ λοιπόν, εσείς βλέπετε να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην ε, τελωνιακή νομοθεσία ή θεωρείτε ότι υπάρχουν περιορισμοί στο εμπόριο ε, ότι ε, δημιουργούνται εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Και τέλος, τελευταία μου ερώτηση. Θυμάμαι ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση Στην περίπτωση επιβολής ε, προστήμων, οποτεδήποτε αυτά καταβάλλονται, επιστρέφονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται με εσά. Φαντάζομαι και εσείς επιβάλλετε πρόστιμα και συγκεντρώνετε χρήματα. Αυτά που διοχετεύονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς ή στο δικό σας προϋπολογισμό ή μήπως σε αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία. Παρακαλώ λοιπόν, έχει το λόγο για να απαντήσετε σε αυτές τις ε, παρατηρήσεις. να απαντήσω στην κυρία Βαϊλέρ για το θέμα των τελωνίων είπατε ότι η Επιτροπή για την Ιστορική Αγορά συνεδρίασε για να εξετάσει τον κοινοτικό τελωνιακό κώδικα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι είμαστε υπέρ της ε, απελευθέρωσης ε, της ροής των εμπορευμάτων έτσι ώστε η εσωτερική αγορά να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Είμαστε υπέρ της ε, διευκόλυνσης του εμπορίου λοιπόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση αυτής της διάταξης με την καταπολέμηση της απάτης. Και έχουμε ένα ελάχιστο ποσοστό προφανώς σε σχέση με όλο ε, όλη τη ροή των εμπορευμάτων που είναι αντικείμενο απάτης. Είναι ελάχιστο το ποσοστό των απατών ε, πραγματικά. Ε, έχουμε πάρα πολύ καλή νομοθεσία, όμως υπάρχει προβλήμα εφαρμογής, υλοποίησης της νομοθεσίας αυτής. Και όταν δηλαδή, πολλές φορές ε, ζητάμε να υπάρξει σωστή διασάφηση, σωστή δήλωση, διαπιστώνουμε ότι λείπουν αρκετά στοιχεία σε κάποιες στήλε. Ενώ μιλάμε για υποχρεωτικέ διασαφήσει. Χωρί αυτέ τι πληροφορίες δεν μπορούμε να εργαστούμε. Και ένα από τα στοιχεία που ανέφερα είναι ότι Τώρα έχουμε κάποιες εταιρείες, Counter Line, οι οποίε κάνουν ε, τη διασάφηση από το Ιράν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν ακολουθεί εξαγωγή προ μία ε, άλλη χώρα της Αφρικής ε, και δεν βλέπουμε ποτέ το όνομα ούτε του πολιτή ούτε του αγοραστή και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα θέλαμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και μιλάμε για ευρωπαϊκές δράσεις δεδομένων που θα επιτρέπουν στην Κομισιό να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ε, τώρα έχουμε πρόσβαση για τη διαμετακόμιση και μπορούμε να έχουμε μια πιο καθολική εικόνα από ότι τα κράτη-μέλη που βλέπουν ένα τμήμα της κίνησης ή όλα εξετάζοντα ε, τι συμβαίνει στη διαμετακόμιση μπορεί να βρει μια μετακίνηση από ένα τελωνίο σε ένα άλλο και μπορούμε να δούμε ε, τις περιπτώσεις όπου υπάρχει απάτη. Αυτές οι πρακτικές φυσικά και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νιούτον για την ε, στήριξή σας όσον αφορά τη συνειδητοποίηση. Η Europol πάντα έτοιμη είναι να βοηθήσει με πρακτικά παραδείγματα ώστε να πετύχει μια εκστρατεία συνειδητοποίηση. Σα ευχαριστούμε πολύ και για την πρόταση που κάνετε για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μα. Θα προωθήσω την ιδέα αυτή στου αρμόδιου. Πάντω, ήδη το κάνουμε σε ένα βαθμό κάθε φορά που υπάρχει μια επιχείρηση ε, παρουσιάζουμε, βάζουμε κάποιες φωτογραφίες για να δείξουμε ότι κοιτάξτε η Europol έχει συνεργαστεί και έχει συντονιστεί με τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη βάζουν κάποιες ταινίες ε, στο YouTube. Το κάνουμε αυτό λοιπόν σε ένα βαθμό. Αυτό που επίσης κάνουμε μερικές φορές κατά την περίοδο των διακοπών μέσω της ιστοσελίδας μας βάζουμε κάποια ανακοίνωση για να βοηθήσουμε και να κάνουμε τους τουρίστες να συνειδητοποιήσουν <clears throat> τι σημαίνει πλαστά προϊόντα και παραποίηση προϊόντων. <clears throat> Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση των ε, υπηρεσιών μας και τις κατασχέσεις αγαθών, σε ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με το Crime Act υπάρχει δυνατότητα ένα ποσοστό της αξίας των κατασχεμένων προϊόντων να πηγαίνει στις υπηρεσίες της αστυνομίας. Δεν γίνεται όμως αυτό σε όλες τις χώρες. Ή συμβαίνει περιστασιακά μόνο. Να πω κάτι για να απαντήσω στην κυρία Βάιλερ ε, για τα πρόστιμα. Υπάρχει μια απόφαση πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των προστιμών στο ποινικό ζήτημα. Έτσι λοιπόν λειτουργεί όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα και αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος μπορούν να εφαρμοστούν τα πρόστιμα και μένουν τα χρήματα αυτά στο κράτος εκεί όπου πρέπει να καταβληθεί το πρόστιμο. Δηλαδή ούτε καν μεταφέρονται τα χρήματα ε, στο κράτος ε, που ζήτησε το πρόστιμο και για την απόφαση πλαίσιο, για την ε, δυνατότητα διασυνοριακής κατάσχεσης και εκεί υπάρχει ένας μηχανισμός κατανομής μεταξύ του κράτου που καταθέτει την αίτηση και του κράτου που προβαίνει στην κατάσχεση. Και πάλι στον ποινικό τομέα. Δεν μιλώ σε διοικητικό επίπεδο, μιλώ για ποινικά ζητήματα. Στον ποινικό τομέα λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά τα χρήματα πηγαίνουν στους εθνικούς προπολογισμού και όχι στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Πριν να ολοκληρώσουμε κάποιες ανακοινώσεις, ε, λοιπόν, στις 2 ε, θα έχουμε στην αίθουσα πολιτός και μια συνέντευξη τύπου όπου θα περιπλεθώ εγώ και ο συγητή και θα υπάρχουν και ορισμένοι εμπειρογνώμονε, ε, κ. Τιεριχέν, κ. Βαστίτκιν, Τζούλια Νόμεν από την Περσία για το Περιβάλλον, ο Στέφαν Στεφάνη από τη Λέγκα Μπιέντη και τον Τσιώτη από τη Λίμπερα. Και να σα πω ότι θα ξεκινήσουμε εμεί εκ νέου τι εργασίε μα στι 3 με θέματα που αφορούν ε, την παρέμβαση της ε, Frontex, ε, του Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Λίμπερα. Θα ξεκινήσουμε στις 3 με το πρώτο πάνελ για την εμπορία ανθρώπων με το σκοπό της σεξουαλικής και της εργασιακής εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Όλαφ, της Europol και της COSI για της παρουσίασής τους και για τη διαθεσιμότητα που δείξατε και φυσικά δείξατε εμπιστοσύνη στις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Εμείς πραγματικά τρέφουμε μεγάλες ελπίδες και είμαστε και πεπισμένοι ότι αυτή η Επιτροπή όταν ολοκληρώσει τη θητεία της, αν και είναι σύντομη θητεία της, θα μπορέσει να εκπονήσει ένα σχέδιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την νομιμοποίηση παράνομων εισόδων. Θα ξανασυναντηθούμε βεβαίως για να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία, αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε στις 3.